Καλησπέρα συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε στην ε, συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας σήμερα το απόγευμα. Έχουμε πολλή δουλειά. Πριν ε, περάσουμε όμως ε, με μια μικρή καθυστέρηση στην ημερησία διάταξη, Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη όπως σας έχει προταθεί. Ωραία, θαυμάσια. Ε, το εκλαμβάνω ως κατάφαση αυτό. Έχουμε διερμηνία από τα Σουηδικά. Ε, θα δούμε ε, αν θα έχουμε και αύριο. Πάντως για σήμερα δεν έχουμε Σουηδικά. Νομίζω καλύπτονται όλοι οι υπόλοιποι γλωσσικός πώς. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, ανακοινώσεις της Προέδρου. Καμία ανακοίνωση δεν έχω. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 24ης Σεπτεμβρίου και της 10ης και 11ης Οκτωβρίου. Έχετε σχόλια για τα πρακτικά? Ούτε. Ωραία. Θαυμάσια. Θα θεωρηθούν λοιπόν εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Which case, I am happy to say, we will move... Οπότε ε, μπορούμε με χαρά να περάσουμε στο πρώτο θέμα για σήμερα που είναι το εργαστήριο με θέμα η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων. Ραδιενεργών δηλαδή. Ε, έχουμε τον δόκτωρ ε, Κλοντ Βαχτέλ που είναι ερευνητής ε, στο Ίδρυμα Στρατηγικής Έρευνας στη Γαλλία και την Ελιζάντε Νέξον που είναι επίσης ερευνητρία στο ίδιο Ίδρυμα και οι Καλοδεχούμενοι και καλωσορίσατε. Θα μας μιλήσετε λοιπόν για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά και πυρηνικά όπλα με ιδιαίτερη έμφαση στους θεσμούς και πώς μπορούμε να ε, ελαχιστοποιήσουμε ή να προλάβουμε τον κίνδυνο για τέτοια ατυχήματα ή συμβάντα ή να αυξήσουμε την αντίστασή μας. Επίσης, ε, περιμένω να ακούσουμε από εσά και τα διάφορα σενάρια προς τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δομές και ικανότητες. Ελπίζω να ακούσουμε και πώς το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμμετέχει περισσότερο στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα όπλα αυτά που εγκρίθηκε πέρσι ε, όταν θα έρθει προς αναθεώρηση του χρόνου για να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε και τι μαθήματα και διδάγματα θα αποκομίσουμε. Ε, θα ήθελα λοιπόν χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Βαχτέλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. <laughs> <laughs> thank you. Je vous remercie, mesdames et Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Εμείς λοιπόν έχουμε επικεντρωθεί στη πιθανή χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο μιας ανταπόκριση σε περίπτωση περιστατικών χημικών, βιολογικών, ιδεολογικών και πυρηνικών όπλων να κάνω μια σύντομη υπενθύμηση για την ε, έκταση των απειλών σε αυτόν τον κλάδο και σε αυτή τη μορφή όπλων μπορεί να είναι και φυσικής ε, προέλευση, όπως επιδημίε και πανδημίες. Για παράδειγμα, έχουμε ε, περιπτώσεις όπως το E. coli, τον έμπολα, ε, που και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια κινητοποίησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και σε κάποια στιγμή θα μπορούσε να έχει φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Έχουμε ε, και ατυχήματα που μπορούν να πλήξουν, για παράδειγμα, χημικές εγκαταστάσεις ή ε, εργαστήρια βιολογικής έρευνας ή με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών που αρχικά μπορούν να προκληθούν από φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, θύελες που μπορεί να προκύψουν από ε, ελληματικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε ε, πυρηνική ακτινοβολία ή εκρήξεις. Ή μπορεί να προκληθούν και από ανθρώπινο σφάλμα, από αμέλεια. Με επικίνδυνες, για παράδειγμα, διαδικασίες ή ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Τέλος, και αυτό που μας ενδιαφέρει μας περισσότερο εδώ, έχουμε τις ε, ε, σκόπιμες ε, πράξεις που μπορεί να προκύψουν από ε, εγκληματικές ενέργειες, ε, τρομοκρατικές ενέργειες, κυρίως ή περιπτώσεις χρήσης που τελικά υποστηρίζονται από κράτη, όπως έχουμε δει τους τελευταίους μήνες. Αυτό μας έχει απασχολήσει. Επομένως, ε, λαμβάνοντα υπόψη ε, την έκταση αυτών των απειλών, η ανακοίνωση του 2009 μαζί με το σχέδιο δράση, ε, επενθύμησε ότι είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της προετοιμασία και ανταπόκριση σε αυτό το πλαίσιο να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για όλες αυτέ τι απειλέ. Γιατί όποια και αν είναι η προέλευση του ενό περιστατικού για ασφα... πολιτικής προστασίας ε, και προστασία της δημόσιας υγείας ε, πρέπει να υπάρχουν κοινέ ενέργειες και προσεγγίσεις παρότι μπορεί να υπάρχουν και μεμονωμένες ε, ενέργειες. Είναι δύσκολο λοιπόν να αξιολογήσουμε αυτέ τι απειλέ, λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε πολύ διαφορετικού κινδύνους, ανάλογα με το περιβάλλον και τη χώρα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η απειλή και μάλιστα αυξάνεται για μια σειρά λόγους. Υπάρχει αρχικά η τεχνολογική ανάπτυξη, ε, υπάρχει το ζήτημα ε, ε, της βιολογικής εξέλιξης σε σχέση με τις απειλές. Διάφορες λοιπόν τεχνολογικές εξελίξεις, στη βιολογική έρευνα, ε, στην υπολογιστική ισχύ και στις μεθόδους ανείχνευσης ε, ε, που μας δυσκολεύουν σε ό,τι αφορά ε, τις τεξουκές ουσίες. Αυτή η απειλή αυξάνεται και επειδή παράλληλα αυξάνεται και η διάδοση των τεχνολογιών αλλά και επειδή έχουμε μεγαλύτερη διάδοση των πληροφοριών που συνδέονται με πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας ε, που είναι πιο ασφαλή απέναντι ε, στην ε, κακοήθη χρήση. Όπως για παράδειγμα για αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουμε στα... κρυπτογράφηση των δεδομένων. Πρέπει να προσθέσουμε και ό,τι έχει να κάνει με την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, η οποία πλέον γίνεται πολύ πιο εύκολα μεταξύ πολλών ε, θεσμών, αλλά μπορεί να αποτελέσει αδυναμία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ό,τι έχει να κάνει και με ε, τους ε, ταξιδιώτες και τα υλικά και άλλα αγαθά. Έχουμε να κάνουμε με τις μεταφορές, ας πούμε, οι εξαγωγές, με σημαντικές ροές και εκεί. Επομένω, ό,τι αφορά την ανάλυση κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντα υπόψη τι πρόσφατε εξελίξει, τι οποίε θα επανέλθουμε σύντομα, έχουμε την χημική απειλή ε, που είναι η πιο μεγάλη από πλευρά ε, σκόπιμης, ε, σκόπιμων ενεργειών. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι πρέπει να προετοιμαστούμε λιγότερο για τους άλλους κινδύνους, κυρίως τους ραδιολογικούς και βιολογικούς. Και εκεί υπάρχει σημαντικός κίνδυνος και θα πρέπει να τα επανεξετάζουμε συστηματικά σε σχέση και με άλλες χώρες για να δούμε τα αποτελέσματά μας. Από την αρχή της δεκαετίας του 2000 λοιπόν είχαμε μία σειρά ε, περιστατικών που συχνά μας επενθυμίζουν ότι πάντα είναι επίκαιρες αυτές οι απειλές. Από το 2010 κυρίως και μετά, σε ό,τι έχει να κάνει, είχαμε και μεγάλα ε, τέτοια περιστατικά, ε, μεγάλες εμβέλειες δηλαδή, όπως ε, στη Φουκουσίμα, παρότι δεν υπήρχε σκόπιμη εκεί. δείχνει όμως τη, το ευάλωτο πολλών από τις εγκαταστάσεις μας. Και εκεί μπαίνει και το ζήτημα της κινητοποίησης στρατιωτικών πόρων σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ε, περίθαλψη των ε, θυμάτων που είτε έχουν δεχθεί εκτινοβολία είτε σε άλλα πλαίσια. Η επιδημία του έμπολα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι ζητήθηκαν στρατιωτικές ενισχύσει και από ΜΚΟ που παραδοσιακά ε, δεν ζητούν τέτοιου είδους ε, βοήθεια και ενίσχυση. Και αυτό μας έδειξε το βαθμό στον οποίο πραγματικά ε, η επιδημία αυτή ξεπέρασε τις δυνατότητες που υπήρχαν και έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη κινητοποίηση. Από τις σκόπιμες τώρα ενέργειες προφανώς έχουμε την χρήση χημικών όπλων και από τους κρατικούς και τους μη κρατικούς φορείς στη Συρία από το 2012 και μετά, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή επικράτεια δηλαδή άμεσα, στο Σάλσμπορι η επίθεση με τον Νόβιτσοκ και δύο ε, απόπειρες οι οποίες ε, απετράπησαν ε, στη Γαλλία και στη Γερμανία και το 2018. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και από τους ε, μη κρατικού φορείς, αλλά και ότι η απειλή που συνδέεται με στήριξη από κρατικού φορείς πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και μάλιστα πολύ σοβαρά. Σε ό,τι έχει να κάνει ε, τα πυρηνικά και ραδιολογικά ε, προϊόντα, βλέπουμε ότι η το λαθρεμπόριο που αποκαλύπτεται συστηματικά, ακόμα κι αν οι στόχοι που αποκαλύφθηκαν δεν ήταν ε, απαραίτητα τρομοκρατικοί, δείχνει όμως ότι υπάρχει ανησυχητική ε, κατάσταση, ότι είμαστε πολύ ευάλωτοι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι σκόπιμε ενέργειε και την ε, χρήση ή τη δυνατότητα χρήση στρατιωτικών ικανοτήτων, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η χρήση αυτών των ε, στρατιωτικών πόρων δεν γίνεται συστηματικά ή αυτόματα, γιατί αφενός ε, ανάλογα με την χώρα τα πάντα έχουν να κάνουν και με τον εθνικό σχεδιασμό. Δεν έχουν όλες αυτές οι χώρες ε, τη δυνατότητα χρήσης στρατιωτικών μέσων. Εξαρτάται και από τον ρόλο των επιμέρους φορέων στη διαχείριση κρίσεων. και αν δεν υπάρχει ε, υπέρβαση των εθνικών δυνατοτήτων μπορεί να μην ε, γίνει χρήση των στρατιωτικών μέσων. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν μια σειρά κριτηρίων θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ταυτοποίηση σενάριων ε, στα οποία θα πρέπει να προστρέξουμε στις στρατιωτικές δυνάμεις και στα εθνικά μέσα μέσω των ε, υπηρεσιών των μυστικών υπηρεσιών, για παράδειγμα, που μπορούσαν να εντοπίσουν ε, μεγάλες ή πολύ σοβαρές απειλές ε, που να αιτιολογήσουν την εκ των προτέρων κινητοποίηση ερωτικών μέσων, για παράδειγμα με μέσα εντοπισμού τέτοιων απειλών. Οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσης, γιατί η κατάσταση αλλάζει πολύ ανάλογα με το αν η κρίση αυτή θα αναπτυχθεί άμεσα και γρήγορα ή αν θα αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου. Ούτε η ανταπόκριση είναι η ίδια. Και για τα στρατιωτικά μέσα αυτό μπορεί να είναι σημαντικό ενδιαφέροντος. Δηλαδή το να γίνει ε, μεσόφρονα τρόπο αυτή η ανάπτυξη των μέσων. Και για τα κράτη-μέλη και για τρίτες χώρες ε, που εμπλέκονται ενδεχομένω. ή πρέπει να δούμε αν το περιστατικό αυτό μπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια για τις ε, εθνικές αρχές και να πρέπει να γίνει χρήση επιπρόσθετων ε, πόρων και μέσων. Επίσης, αν υπάρχει ε, επανάληψη στο χρόνο ή και ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των περιστατικών, αν γίνεται έτσι κατακρεματισμένα εξελίσσεται τη κρίση. Μεταξύ των κριτηρίων έχουμε και την δυνατότητα των ε, κρατών μελών να ανταποκριθούν με την ενίσχυση ε, του προσωπικού του των αξιωματούχων τους, όταν αυτοί ε, κινητοποιούνται κάπου αλλού ή όταν υπάρχει δυνατότητα ε, χρήσης ε, εξειδικευμένων μονάδων με πολύ ειδικέ ε, δυνατότητες και ικανότητε. ή κατά πόσο το προσωπικό είναι καλά εκπαιδευμένο ε, για να παράσχει, για παράδειγμα, πρώτε βοήθειες ε, σε ό,τι αφορά την θύματα σε συγκεκριμένε περιπτώσεις και απειλέ. Το τελευταίο. Άλλες μορφές και κατηγορίες συμφωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα, διμερεί συμφωνίε συνεργασία όταν έχουμε διασυνοριακή απειλή ή κινητοποίηση, κινητοποίηση και χρήση συμφωνιών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έχουμε εντοπίσει μια σειρά σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην χρήση στρατιωτικών μέσων. Έχουμε την εκ των προτέρων πρόληψη, Μπορεί να γίνει χρήση αυτών των μέσων λοιπόν για την ενίσχυση σε ε, προσπάθειες αύξηση των ικανοτήτων ε, και σε τρίτες χώρε για να υπάρχει ένα συνεχέ μεταξύ ασφάλεια στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό. Οι ε, στρατιωτικέ επιχειρήσει μικρή κλίμακα και άμεση ανάπτυξη, που μπορούν να επιτρέψουν την παρέμβαση σε συγκεκριμένε κρίσει όταν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος ροπή και πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Το δεύτερο σενάριο. Επίθεση ή καταστροφή μεγάλης κλίμακας ε, που υπερβαίνει τις ε, δυνατότητες ανταπόκρισης ε, του κράτους μέλους ή των κρατών μελών ή όταν έχουμε μία συνεχιζόμενη απειλή ή επαναλαμβανόμενες απειλές ε, που πάλι ε, δοκιμάζουν ε, τις δυνατότητές μας. Ένα σενάριο το οποίο απαιτεί την χρήση εξειδικευμένων δυνατοτήτων ή δυνατοτήτων εχμής που συχνά έχουν στρατιωτικές δυνάμεις Βλέπουμε για παράδειγμα τις δυνατότητες παρέμβασης σε περιβάλλον ε, όπου υπάρχει ε, ραδιενέργεια. Δυνατότητες όμως που ε, απαιτούν συστηματική κατάρτιση και επανεκπαίδευση για παράδειγμα στην απομόλυνση. Εκεί υπάρχει ε, πρόβλημα ενδεχομένω γιατί δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο αυτό από τα κράτη. Ή και στον ιατρικό τομέα αντίστοιχα, στον τομέα της περίθαλψη. Ένα άλλο σενάριο, έχουμε την χρήση βιολογικών ε, και χημικών ε, ουσιών στρατιωτικού χαρακτήρα και εκεί μπορεί να υπάρξει υποψία εμπλοκής ενός κράτους μετά, υβριδική απειλή με πτυχή χημικών, βιολογικών, βιολογικών και πυρονικών όπλων και έχουμε την ε, σύγκληση και διασύνδεση διαφόρων στοιχείων όπου τελικά μας οδηγούν σε μία πολυδιάστατη και πιο πολύπλοκη απειλή ε, κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ε, κρίσιμης σημασίας σε εγκαταστάσεις και υποδομές. Εδώ η ανταπόκριση θα μπορούσε να αφορά την ασφάλεια μας ε, και την ανταπόκριση ως προς ε, την κυβερνοεπίθεση και όχι προς τα χημικά και άλλα όπλα. Τέλος, κάτι άλλο το οποίο είναι ε, πιο ακραίο έχει να κάνει με τις ε, συνέπειες που προκύπτουν από έναν πόλεμο ή μια σύγκρουση. Πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πιο ευνοϊκά προς ε, την επιθανή ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων σε περίπτωση κρίσης. Αφενός έχουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει πολλάκις κατοχυρωθεί ε, και σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολιτικές δηλώσεις εκπροσώπων των κρατών μελών με ακρογωνιαίο λίθο την ε, στρατηγική του 2016 που υπενθυμίζει ότι η φιλοδοξία της στρατιωτικής αυτονομίας ε, εξακολουθεί να ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν εκκλήσεις ε, για την ασφάλεια και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρονται οι απόπειρε ή προσπάθειε μάλλον για την ε, άμυνα, αλλά και το έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Καλούνται επίση τα κράτη-μέλη να πράξουν τα δέοντα, ούτω ώστε η προσήλωσή τους αυτή να μεταφράζεται πλέον και σε ενέργειες. Όλοι αυτοί είναι τρόποι βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ δηλώσει, και πολύ πρόσφατα μάλιστα είχαμε αυτή του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, το Νοέμβριο του 2018, πριν από μερικέ μέρε, ε, σε ό,τι φορά μετά, μάλλον κατά την εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 ετών από, τον, ε, από, τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου τα κράτη-μέλη ε, να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης. Και η κυρία Μέρκελ, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ολομέλεια λοιπόν του Νοεμβρίου, μίλησε για ένα όραμα, ώστε μία μέρα να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό. En Έχουν αλλάξει λοιπόν τα πράγματα, αλλά έχουμε αντίστοιχα και πολύ σημαντικές εξελίξεις από το 2016-2017 Πρώτα απ' όλα, η μόνιμη ε, διαρθρωμένη συνεργασία, ΠΕΣΚΟ, με απόφαση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017, που με θελοντικό τρόπο όμως εμπλέκει την πλειονότητα των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία. Μπορούμε να μιλήσουμε και για την ε, ε, κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας αυτό συνδέεται και με άλλες πρωτοβουλίες άμυνας και υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Εξωτερικής, δράση και από τον EUMS και από την EDA. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στον τομέα που μας ενδιαφέρει εδώ σήμερα. Σε το πλαίσιο λοιπόν ε, τη μόνιμη διαρθρωμένη ε, συνεργασία ε, ξεκίνησαν μια σειρά project από τις αρχές του 2018. Κανένα δεν αφορά συγκεκριμένα τα χημικά, βιολογικά και άλλα όπλα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική στήριξη που θα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε σε περίπτωση κρίση. Κάθε χρόνο επιλέγονται και άλλα έργα, άλλα project, οπότε υπάρχει δυνατότητα να επιλεγεί συγκεκριμένα ένα τέτοιο project, ε, NRBC. Για παράδειγμα, είχαμε ένα τέτοιο project για την Κεντρική Ευρώπη, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ε, συστήματος εποπτείας, ε, ροπή, που να δώσει έμφαση στις επιχειρησιακές πτυχές σε ό,τι έχει να κάνει και με τη θάλασσα. άλλη πρωτοβουλία είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης που διακρίνει μεταξύ της ε, ΠΕΣΚΟ και ξεκίνησε από τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο, με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας. Συμπληρωματικά λειτουργεί βέβαια σε σχέση με την άμυνα στην Ευρώπη και σε επίπεδο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να το δούμε σαν τη διαστολή δηλαδή με τα υπάρχοντα μέσα. Και έχει λάβει τη στήριξη 9 Υπουργών Άμυνα ε, τον Ιούνιο του 2018. Έχουμε λοιπόν ω στόχο ένα κοινό σχεδιασμό άμυνα, ούτω ώστε ε, να ενισχύσουμε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγέ ε, προσωπικού και κοινέ ασκήσεις με συνεργασία μεταξύ χωρών που έχουν την πολιτική βούληση να ενεργήσουν από κοινού και την στρατητική ικανότητα να το πράξουν σε διάφορα σενάρια. Το οποίο δεν έχει μόνο στρατηγική χρειά, αλλά και πολιτική. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εδώ. Για παράδειγμα, έχουμε Βρετανική και Ολλανδική παρέμβαση στην Καραϊβική, που μπορεί να αιτιολογήσει την, ε, μια τέτοια πρωτοβουλία στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας ε, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο σχέδιο δράσης NRBC του 2018 ζητούσε στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικών εταίρων. Αυτό σαφώς ε, και περιλαμβάνει και το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια πρέπει να αναπτύξει τις ε, ικανότητές τη. Αυτό θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά ως προ τα όσα γίνονται σε επίπεδο ΝΑΤΟ και να μην έρχονται όλα αυτά σε αντιδιαστολή. Η κοινή διακήρυξη για τις δυνατότητες συνεργασίες στην Σύνοδο ε, του ΝΑΤΟ του 2016 και είχαμε και μια ε, νέα κοινή δήλωση στο πλαίσιο ή μάλλον εν ώψη της Συνόδου Ακορυφής των ΝΑΤΟ τον Ιούλιο του 2018 με στόχο την ενίσχυση της ε, ανθεκτικότητας απέναντι σε απειλές ε, σε χημικά, βιολογικά, ροδιολογικά και πυρηνικά όπλα. Μίλησαμε λοιπόν για συνεργασία σε επίπεδο προσωπικού μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για την προετοιμασία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνων, σε ό,τι αφορά την ιατρική παρέμβαση ε, την ανταπόκριση σε περιστατικά μεγάλης εμβέλεια ε, και ούτω καθεξής. Μπορούμε να υπερθυμίσουμε την πρόσφατη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών, Πολλά κατημέλη συμμετέχουν εκεί, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε περαιτέρω προσπάθειες για την βελτίωση της ανταπόκρισης με κοινέ ε, ε, ασκήσεις, συζητήσεις και το καθεξής. Και ο τομέας NRBC ε, είναι από αυτούς που έχουν αναφερθεί ρητός ως σημεία ενδιαφέροντος και τομείς ενδιαφέροντος για αυτό το κέντρο αριστείας. Είναι χρήσιμο να προσδιορίσουμε καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ επιμέρους κέντρων κρίσεων που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό όπως η Europol και, έχουν, και εξαρτώνται από την Επιτροπή ε, Κρίσεων του ΝΑΤΟ όπως ε, η Emergency Planning Committee. Τέλος, και γενικώ πώς έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασία, ε, που είναι θεμέλιο όλης αυτής της ευρωπαϊκής ανταπόκριση Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού ε, Ανταπόκρισης σε έκτακτες περιστάσεις, το ERCC. Και το ERC ε, που συγκεντρώνει επιμέρους μέσα και πόρους των κρατών μελών. Και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα που εντάσσεται στο ERC σε περίπτωση κρίσεων όλα αυτά βέβαια προς το παρόν μένουν λίγο θεωρητικά ε, και δεν είναι πάντα διαθέσιμα γιατί μπορούν, μπορεί να τα χρειαζόμαστε κάπου αλλού. Γι' αυτό είναι μικρό το κίνητρο ε, για τα κρατημέλη να δώσουν πόρους εκεί γιατί αυτή τη στιγμή ε, τα επιχειρησιακά κόστη δεν χρηματοδοτούνται και είναι και τα περισσότερα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει ειδικό αποθεματικό για την πολιτική προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να χρησιμοποιείται βέβαια σε, σαν έσχατη λύση, αλλά να είναι πάντα διαθέσιμο και να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να ε, αποφασίζεται έτσι η κινητοποίηση του μηχανισμού και η κατανομή που μπορεί να οδηγήσει σε διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων. Πρέπει βέβαια να θεσπιστεί και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γνώσεων ε, στον τομέα της, ε, προστασίας, της πολιτικής προστασίας. Οι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυάριθμε σε ό,τι αφορά την ε, πρόληψη αυτών των περιστατικών μεγάλη κλίμακα στον τομέα των χημικών, βιολογικών και άλλων όπλων, με έλεγχο στι εξαγωγέ, προστασία των κρίσιμων υποδομών, στήριξη προ διεθνεί οργανισμού, όπω ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ή προστασία από τα χημικά όπλα, πολύ σημαντικέ ε, προσπάθειε για τη χρηματοδότηση τη έρευνα και ανάπτυξη. είτε με κοινά ερευνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με, στο πρόγραμμα Ορίζον 2020, είτε αλλού προγράμματα ε, προειδοποίησης, έγκαιρης προειδοποίησης σε ό,τι αφορά τις ε, μεταδοτικές ασθένειες, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων, ε, στο πλαίσιο, για παράδειγμα, συνεργασίας ε, στον ορίζοντα 2020, χρηματοδότηση χρηματοδότηση ασκήσεων, ενίσχυση της ποινικοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών, κάτι το οποίο έχει γίνει τελευταία. Δυνατότητα ανταλλαγής ε, μυστικών πληροφοριών ε, μεταξύ κρατών μελών ή τελικά δυνατότητα περιορισμού ε, της παράνομης διακίνησης υλικού NRBC με τρίτες χώρες. Εδώ βλέπετε λοιπόν έναν ε, μη πλήρη κατάλογο για να σας δώσω μια εικόνα της έκτασης όμως ε, των ευρωπαϊκών προσπαθειών στον τομέα της πρόληψης. Ο συντονισμός σε περίπτωση κρίσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ θα προσθεθούν και στρατιωτικά μέσα. Είναι περίπλοκο βέβαια το ζήτημα γιατί έχουμε μια πλειάδα ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών και μέσων που κινητοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Έχουμε και τα κράτη-μέλη, την, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης, ε, του επιμέρου ε, φορεί Ευρωπαϊκής Ένωσης, Europol, Eurojust. Να μην τα αναφέρω τώρα όλα διεξοδικά. Και εμπειρογνώμονε των κρατών μελών ή διεθνών οργανισμών όπως ο ΠΟΗ. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Έχουμε λοιπόν ε, πολλούς και διαφορετικούς φορείς και είναι σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός συντονισμού. Έχουμε το IPCR για την ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσεων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας πιο ευέλικτος μηχανισμός που έχει συσταθεί από το 2013 και επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και μέσων σε περίπτωση κρίσης και ενεργοποιείται αυτόματα όταν ένα κράτος μέλος ε, ε, επικληθεί την ρήτρα αλληλεγγύης. Και τώρα, περισσότερο για τα στρατιωτικά μέσα και ικανότητε, να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο και περιβάλλον που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί έτσι πολλές προκλήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την προσάρτηση της ε, Ουκρανίας από τη Ρωσία το 2014, αλλά Έχουμε και ενίσχυση ε, των πολιτικών συγκεκριμένων κρατών μελών μετά και από τρομοκρατικές απειλές ε, που διαδέχονται μία την άλλη στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και είναι φύσεως ε, τέτοιας. Και μετά έχουμε και την στάση της αμερικανικής πλευράς για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ και πώς αυτό συνδέεται και με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ε, στήριξη των ε, πολυμερών συμφωνιών για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με τις προεκτάσεις και συνέπειες του Brexit. ενώ παλαιότερα οι σύνδεσμοί μας με το ΝΑΤΟ και η ευρωπαϊκή ανταπόκριση ήταν πιο δύσκολο να τα αναφέρουμε, να αναφερθούν. Ευχαριστώ. Thank you, And... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Βάχτελ. Ε, έχουμε άλλα 20-25 λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Λοιπόν, ποιο είναι το πλαίσιο αυτής της δυνατότητας ε, ε, επίκλησης ε, και χρήσης στρατιωτικών μέσων σε επίλυση κρίσεων NRBC. Αρχικά έχουμε την σφαιρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2016 και μετά την στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας του 2015. Είναι λοιπόν δύο σφαιρικά κείμενα που δεν υπησέρχονται σε λεπτομέρειες ότι αφορούν τα NRBC όπλα, αλλά ισχύουν και για αυτά. Οι αρχές που βρίσκονται στην βάση αυτής της στρατηγικής είναι ότι ε, το κράτος μέλος, ε, το ενδιαφερόμενο, έχει την βασική ευθύνη για την επίλυση της κρίσης και τη διαχείριση της κρίσης στην επικρατειά του, αλλά αναγνωρίζεται ότι οι απειλές CBRN είναι περίπλοκες, είναι δύσκολο να επιληθούν και έτσι μπορούμε ενδέχεται να υπάρξει υπέρβαση των μέσων του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και γι' αυτό αιτιολογείται και ε, η επίκληση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Η ρήτρα αμυσαίας συνδρομής, άμυνας, και αλληλεγγύης των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αρρωγή, υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Για να επικληθεί ένα κράτος μέλος αυτή τη ρήτρα, πρέπει αρχικά να αντιμετωπίζει μία ένοπλη επίθεση θα δούμε όμως ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ε, σφαιρικά αν θέλετε και ότι η επίθεση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στην επικράτειά του. Είναι μια ρήτρα που είχε ζητήσει ο Γάλλος πρόεδρος ακριβώς μετά τις επιθέσεις ε, στη Γαλλία τον Νοέμβριο του 2015. Η αποστολές που προκύπτουν από αυτή την ρήτρα έχουν πολλές μορφές. Συμπεριλαμβάνουμε και τις κοινέ δράσεις ε, για τον παροπλισμό, ε, ανθρωπιστικές ε, ενέργειες διάσωσης, αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από ε, ε, μεγάλες φυσικές καταστροφές, ε, αποστολές πρόληψης και αποφυγής συγκρούσεων, και επιχειρήσεις, αποκατάσταση της ειρήνης, σταθεροποίησης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο άρθρο 43 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βέβαια έχουμε και τον ρόλο της ε, πολιτικής προστασίας και του στρατικού σκέλους. Και σε αυτό το σταυροδρόμι λοιπόν βρισκόμαστε και βλέπουμε την ιδιαιτερότητα της στρατιωτικής παρέμβασης στην πλειονότητα των περιπτώσεων στο πλαίσιο της Ένωσης. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτών των ε, μέσων θα γίνεται όταν έχουμε, βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι μεταξύ πολιτικής προστασίας και στρατιωτικού σκέλους. Με το πιο συμβατικό τρόπο. Είπα λοιπόν ότι η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή ε, έχει ορισμένε προποθέσει. Υπάρχει και η ρήτρα αλληλεγγύη από την άλλη. Υπερθυμίζω ότι είναι αρκετά ιδιαίτερη γιατί προβλέπει το ετών κράτος μέλος, το ετούν κράτος μέλος να έχει ε, εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που του προσφέρονται για να επιληθεί αφενός η κρίση και ότι υπάρχει υπέρβαση αυτών των δυνατοτήτων αφετέρου. Μίλησα για την έκκληση της Γαλλίας που είχε γίνει, στην, που συμπεριλήφθη στην ρήτρα ε, συνδρομής. Δεν βρισκόμαστε σε περίπτωση υπέρβασης των ε, εθνικών μέσων, παρότι ήταν ε, πολύ μεγάλο το τίμημα αυτή τη τρομοκρατική ενέργεια. Όμω, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιπτώσει ενισχυμένη συνεργασία με ευρωπαϊκέ χώρε σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγμα, για να υπάρξει άμεση ε, ανταπόκριση για την ε, εξουδετέρωση των τρομοκρατών, όπως συνέβη ε, και στην περίπτωση της Γαλλία. Alors, euh, en ce qui concerne Euh, les euh, euh, en ce qui concerne Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσταθέμενη αξία της χρήσης στρατητικών μέσων, έχουμε μία σειρά παραδείγματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Δεν είναι κάτι το καινούριο λοιπόν. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η επιδημία έμπολα του 2014, όπου είδαμε αρχικά την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είχαμε μια νέα και αξιοσημείωτη ε, συμφωνία και μετά είδαμε ποια θα μπορούσε να είναι συμβολή των στρατιωτικών μέσων σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε μεγάλο βαθμό η παρέμβαση και αντιμετώπιση έγινε από ΜΚΟ, παρότι στην πορεία προέκυψαν περίπλοκα ζητήματα και εκεί τα στρατιωτικά μέσα, οι στρατιωτικές δυνάμεις με την εξειδικευμένη τους γνώση, ε, τα εξειδικευμένα τους μέσα, ιατρικής παρέμβαση και άλλη. Στη Γαλλία ήταν η αντίστοιχη υπηρεσία στρατιωτικής ιατρικής ε, που κατάφεραν να δημιουργήσουν εξειδικευμένα κέντρα περίθαλψης των θυμάτων γιατί αυτά τα θύματα έπρεπε να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργήθηκαν ε, εκεί με ικανότητες, ε, στρατηγικές ικανότητες εχμής. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι κάτι που απασχολούν και τις στρατιωτικές περιπόλους, οι οποίες περιπολούν για την ασφάλεια ορισμένων εγκαταστάσεων. Έχουμε δει και εδώ στις Βρυξέλλες, ε, σήμερα το πρωί που φτάναμε, είδαμε μια τέτοια περίπολο. Ε, συμμετέχει λοιπόν και ο στρατός, ε, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τρομοκρατικής φύσεως, που κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι πολιτικό, όχι στρατιωτικό σκέλος. Ε, έδωσε και όλο το παράδειγμα για τον κυκλώνα Ήρμα και τις ε, αρμοδιότητες, όπου έχουμε πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα. Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Νόβιτσοκ, που χρησιμοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και το Πολώνιο 210 πριν από λίγα χρόνια, όπου ε, υπάρχουν ιδιαικές αρμοδιότητες Ε, του στρατού και χρησιμοποιήθηκαν ε, για, ως πραγματογνωμοσύνη δηλαδή κυρίως και για τη διερεύνηση ε, χρήσης όπλων χημικών, βιολογικών και βιολογικών και πυρηνικών γιατί αυτά είναι ευρύτερα γνωστά στο στρατιωτικό τομέα και λιγότερο στους πολίτες. Ποια είναι τώρα τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ε, ε, για τη χρήση στρατιωτικών μέσων για να αντιμετωπίσουν κατεπίγουσες καταστάσεις πολιτικού χαρακτήρα. Πολύ συχνά αυτό συνδέονται με το εξής. Τα στρατιωτικά μέσα και οι στρατιωτικοί δεν είναι συνηθισμένοι πάντα να συνεργάζονται με τις ε, πολιτικές υπηρεσίες και πόσο μάλλον να είναι υπό τις διαταγές ε, κάποιου πολιτικού προσωπικού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αρμοδιότητες και ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν και να προαχθεί η συνεργασία. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι οι ε, βασικές δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και κυρίως ε, ε, μια ανάγκη πάρα πολύ σφοδρή για τα χημικά, βιολογικά και ραδιολογικά όπλα. Είναι ιδιαίτερα τεχνικό και θα πρέπει να προετοιμάζεται η δουλειά αυτή και να προγραμματίζεται σε συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών μέσων. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα παντού και θα πρέπει να προετοιμαστεί και να ασκηθεί επιτόπου, να γίνονται δηλαδή αντίστοιχε ασκήσεις και γυμνάσια και προετοιμασίες. Στη συνέχεια υπάρχει ε, όντως η οργάνωση ε, της ε, ε, και της ιεραρχίας και πώς συνδέεται αυτό και συντονίζεται ο στρατός με τους πολιτικούς φορείς. Ε, και αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμάζεται σε επίπεδο επιτελείων. Κάτι άλλο που είναι επίσης δύσκολο, στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ο επιμερισμός των ε, αρμοδιοτήτων δεν είναι πάντα ο ίδιος. Ας πούμε, δεν έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες, οι πυροσβέστες, η αστυνομία, οι δυνάμεις ε, ασφαλείας, ε, οι ιατρικοί ε, φορείς και σώματα δεν έχουν παντού τις ίδιες αρμοδιότητες σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί η αποστολή του καθενός και τα καθήκοντά του και μάλιστα ε, όταν ε, συμμετέχουν σε μία παρέμβαση, σε μία επέμβαση διάφορες δυνάμεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει ο καθένας να γνωρίζει τις αρμοδιότητές του. Άλλο σημαντικό είναι η θεώρηση που έχει κάθε χώρα για το ρόλο των στρατιωτικών μέσων που μπορεί να αναπτύξει. Σε πολλές χώρες τα στρατιωτικά μέσα είναι εσχά της καταφυγής όταν πραγματικά δεν αρκούν τα πολιτικά μέσα για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το κοιτάξουμε, αλλά υπάρχουν και κάποιες χώρες για τις οποίες η στρατιωτική επέμβαση είναι κάτι το συνηθισμένο, ας πούμε, σύνηθες και θεσμοθετημένο ως ε, συμπληρωματικό σε περίπτωση σημαντικής θεομηνίας. Ε, ε, ε, καταστροφής. Για παράδειγμα, στη Γαλλία έχουμε στρατιωτικά μέσα τα οποία μονίμως είναι στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών. Αλλά και εκεί κάθε χώρα έχει τον τρόπο που λειτουργεί και τη φόρμουλα η Αυστρία έχει καταθέσει σχετικά μια μελέτη που έχει γίνει, αλλά και άλλες χώρες ε, προβληματίζονται για τα συγκεκριμένα θέματα και για το ρόλο, το θεσμικό ρόλο ε, του στρατού και ποιος ε, θα είναι αυτός ο ρόλος απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές και σε ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. κάτι άλλο που δεν είναι τόσο δυσκολία όσο πρόκληση. Και αν υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα ε, στα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά όπλα, το 2017 είναι ό,τι έχει να κάνει με την επεμβάσεις, με τη διαλειτουργικότητα για το πώς μπορεί ο στρατός να συνεργαστεί με τα, την πολιτική προστασία έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές και αυτά τα προβλήματα. Ας πούμε, αν χρειαστεί μια μονάδα που εργάζεται στην από μόλυνση των θυμάτων να αντικατασταθεί, γιατί στέλνουν αυτή τη μονάδα σε ένα άλλο κράτος μέλος, ε, να μπορεί αυτή να αντικαθίσταται ε, από άλλη υπηρεσία χωρίς να έχει πολύ διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ε, γιατί μπορεί να προέρχεται από άλλη χώρα. Αυτό μπορεί να χρειάζεται και ενίσχυση ως προς τον εξοπλισμό και τον υλικοτεχνικό και την εξάρτηση που έχουν τις στολές. Ε, ένας άλλος ρόλος, τον οποίο θα μπορούσε κανείς να ε, δώσει στο στρατό, να επιφορτήσει το στρατό ανάλογα με τις ιδιαιτερότητά του εκ των προτέρων, είναι η συνεισφορά ε, στις πληροφορίες και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Πολύ σημαντικό. για να έχουμε πολύ στοχευμένη απάντηση. με ε, ενδεχομένως συμμετοχή στρατιωτικών μέσων. Επίσης, εκ των προτέρων, είναι μια δουλειά που γίνεται για την έρευνα και την ανάπτυξη για πιο ε, αποτελεσματική απόκριση ε, στην τρομοκρατία τύπου χημικού, βιολογικού, ραδιολογικού ή πυρηνικού. Εκεί μπορεί να δοθούν οι αρμοδιότητες αυτές από τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό. Κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η άσκηση και οι κοινέ ασκήσεις και τα γυμνάσια των διαφόρων ε, υπηρεσιών στρατιωτικών και πολιτικών. Κοινέ πάντα προσπάθειες και ασκήσεις και στα διάφορα ε, ευρωπαϊκά κράτη για να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κατάσταση η πρώτη τέτοια άσκηση, οι πρώτες τέτοιες ασκήσεις ήταν κυρίως ασκήσεις ε, επίδειξης κοινή, δηλαδή όπου κάθε χώρα έδειχνε στην άλλη πώς λύνει τα προβλήματα. Όπως στην απομόλυνση ε, μια τέτοιας ε, ε, επίθεσης, ε, πέρα από την επίδειξη λοιπόν, τώρα θα πρέπει να περάσουμε και σε ασκήσεις επιχειρησιακές, έτσι πιο περίπλοκες και πιο ε, εξελιγμένες, για να δούμε πώς μπορεί ας να δίνει τη σκητάλη η, μια μονάδα από μια χώρα μέλος, μια άλλη από μια άλλη χώρα ε, μέλος. Επίσης, κάποια παραδείγματα ε, ε, από καταστάσεις κρίσεων θα σας έδινα γρήγορα για τους στρατούς, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει η δημιουργία μιας ε, ζώνης αποκλεισμού. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια χημική επίθεση τρομοκρατική, έχουμε ένα κλειό στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος οποιονδήποτε δεν έχει συγκεκριμένη ε, στολή, ε, εξοπλισμό και αποστολή και ρόλο στο συγκεκριμένο κύκλο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ε, επιχείρηση, δύσκολη σε αστικό περιβάλλον και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύτιμο αν έχει κανείς πολύ γρήγορα ενισχύσεις. Γιατί οι πολιτικές μονάδες και ομάδες που δεν είναι συνηθισμένες ε, να έχουν μια έντονη σωματική δραστηριότητα με προστατευτικές στολές, τρεις και τέσσερις ώρες. Άρα θα μπορούσε να ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή μια ομάδα από τη χώρα στην οποία έγινε η επίθεση, αλλά στη συνέχεια να συμμετέχει και ο στρατός ενδεχομένως και από όλη χώρα. Το ίδιο πλεονέκτημα υπάρχει και με ε, όλη τη γνώση που έχουν οι στρατιωτικοί γιατροί που δεν είναι η μόνη, είναι σχεδόν η μόνη ε, που έχει τέτοιες αρμοδιότητες και γνώσεις για ε, ε, τοξικολογικές πολεμικές επιθέσεις, είτε μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε μετά από, από, από, μόλυνση πολύ επιθετικών ραδιενεργών στοιχείων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και όλη η φάση μετά την κρίση, η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική. για την ιατρική παρακολούθηση και περίθρεψη των θυμάτων. Ιδιαίτερα όταν είναι χημικά τα όπλα, έπαιρνανε μήνες ολόκληρους στο νοσοκομείο. Είδαμε μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, πολλές ε, χώρες και η δική μου δέχτηκαν ε, θύματα που είχαν υποστεί ε, επίθεση με χημικό αέριο, υπερίτη, ε, και ήταν πολύ μακροχρόνια η θεραπεία και αποθεραπεία. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τέτοια γνώση, η γνώση αυτή κυρίως προέρχεται από το στρατό. Δηλαδή, αν έχουμε κάπου 100 θύματα ε, ε, από υπερίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα πρέπει να μοιραστούν οι χώρες μέλη τα θύματα αυτά γιατί κάθε ένα από τα θύματα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Επίσης, οι δυνατότητες έρευνας που αφορούν ε, και πάλι τους παράγοντες πολέμου ακόμα και αν είναι τρομοκρατική επίθεση και είναι πολιτική προστασία, ο στρατός έχει ιδιαίτερη γνώση για τέτοιες ε, πολεμικού τύπου επιθέσεις. Μετά από όλα αυτά, λοιπόν, ε, για να δούμε ποιοι είναι οι προσανατολισμοί. Ε, les σημαντικότεροι τουλάχιστον προσανατολισμοί που θα μπορούσαμε να δώσουμε ως συμπεράσματα. Θα πρέπει τα διάφορα κράτη-μέλη από κοινού να κοιτάξουν τα διάφορα σενάρια που μπορεί να προκύψουν και να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι που από κοινού θα πρέπει να εξυπηρετηθούν αν υπάρχει ας πούμε βρώμικη βόμβα που ε, ε, διαδίδει ένα ραδιενεργό στοιχείο ή μια χημική επίθεση με μια χημική ουσία. με υπερήτη αερομουστάρδας και τα λοιπά που διαχέεται ε, στο περιβάλλον ή ακόμα και βιολογικό όπλο ένα μικρόβιο, ένας παθογόνος ε, παράγοντας, πολύ μολυσματικός. Ε, αυτή η δουλειά θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία μεταξύ των διαφορών κρατών μελών και χρειάζεται κοινή ε, προσπάθεια προγραμματισμού για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος κάθε υπηρεσίας και να γνωρίζει κάθε χώρα πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης οι εξοπλισμοί και οι δυνατότητες να προσαρμόζονται, να υπάρχει και συντονισμός και συνεργασία ε, για τις ασκήσεις και την εκπαίδευση του προσωπικού. Une, ε, en Τώρα, ως προς την οργάνωση, ε, ένα πρώτο στάδιο και μια δυνατότητα θα ήταν να σκεφτούμε ένα σύστημα σε δύο επίπεδα. Όπως ε, ε, αυτά που προτείνονται στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Ε, θα μπορούσαν οι διάφοροι στρατοί να έχουν αντίστοιχες μονάδες στους τομείς όπου ειδικεύονται και όπου η αρμοδιότητα είναι κυρίως στρατιωτική περισσότερο και λιγότερο πολιτική. Euh, euh, euh, λοιπόν, ένα δεύτερο ε, που θα μπορούσε να προτείνει κανείς ε, υπάρχουν κάποιες μονάδες που έχουν λίγο προσωπικό αλλά πάρα πολύ εξειδικευμένο. Ε, αυτό θα μπορούσε να ε, οδηγήσει στη δημιουργία μιας κοινή εφεδρείας κυρίως ως προς το υλικό και τον εξοπλισμό όπως γίνεται και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και θα ήταν συμπληρωματικό εκεί που είναι πολύ ανεπτυγμένη η πραγματογνωμοσύνη στα στρατιωτικά και ένα δεύτερο επίπεδο πέρα από το τεχνικό θα ήταν να υπάρχει σε ένα δεύτερο επίπεδο, ένα προσωπικό ίσως λιγότερο ειδικευμένο, αλλά αυτή τη στιγμή εξαντλήσει η χώρα στην οποία έγινε η επίθεση ε, τις εφεδρίες της που έχει σε προσωπικό, να πάρει τη σκητάλη άλλη χώρα και να ενισχύσει ε, σε προσωπικό ε, την αποστολή αυτή. Για τις πρωτοβουλίες, να τελειώνω, που είναι πρωτοβουλίες περισσότερο ανάληψης ευθυνών ή αποστολών που αξίζει να μελετηθούν ως προς την εφικτό, το εφικτό τους και που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα σημερινά προγράμματα για τα πυρηνικά, χημικά, ραδιολογικά και πυρηνικά είναι να υπάρχει διαβούλευση στα διάφορα κράτη-μέλη να ρωτήσουμε πώς βλέπει κάθε χώρα το ρόλο της για τη συμμετοχή στρατιωτικών μέσων. Ποια είναι τα στρατιωτικά μέσα που θα μπορούσε η κάθε χώρα να διαθέσει, ε, σε ποιες ε, συνθήκες και στη συνέχεια... επειδή θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό δόγμα επέμβασης για να υπάρχει αυτή η διαλειτουργικότητα, Ίσως να έπρεπε να αρχίσουμε από κάτι που θα έμοιαζε με ένα συμπόσιο ε, που θα συνεδριάσουν ε, και θα διαβουλευθούν οι ειδικοί από τα διάφορα κράτη-μέλη ως προς το εκάστοτε δόγμα που έχει κάθε χώρα παρέμβασης και επέμβασης και πώς θα μπορούσαν να ε, συμπλησιάσουν τις διάφορες αυτές δράσεις ή τουλάχιστον το βασικό κορμό, το σκελετό, για να μπορούν να συνδράμουν και οι άλλες χώρες για μια αλληλο βοήθεια. Με απότερο στόχο να υπάρχει ένα κοινό αποθεματικό, μια εφεδρεία υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε Ευρώπη, όχι μόνο με πολιτικά μέσα αλλά και με ορισμένα στρατιωτικά μέσα που μπορεί πολύ γρήγορα να πηγαίνουν όπου χρειάζεται, όπου έχει γίνει μια επίθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Dr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βάχτελ και φαντάζομαι θα υπάρξουν αρκετές ε, ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Ένας τουλάχιστον ε, συνάδελφος έχει ήδη πει ότι θα ήθελε να μιλήσει. Ο κύριος Γκάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση που είχατε. Μας δώσατε έτσι μια γενική εικόνα και βεβαίως εγώ ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τελικά, όταν προκύπτει ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο είναι σημαντικό, Υπάρχουν ε, άλλες δυνατότητες ε, δοκιμών επιχειρήσεων που να μπορούν να λάβουν χώρα από πλευρά αρμόδιων αρχών. Δηλαδή, έχετε έτσι μια γενική εικόνα για τα διάφορα κράτη-μέλη, κατά πόσον διεξάγονται δοκιμές, κατά πόσο ενδεχομένω να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι και πέρα από τα σύνορα μίας και μόνο χώρας. Δηλαδή, γνωρίζουν οι Βρυξέλλες ποιος έχει τι τι είναι διαθέσιμο και τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ή μήπως εξακολουθείτε να βρίσκεστε έτσι σε κάποια πολύ αρχική φάση. Δηλαδή πρώτα ενημερώνεται κανείς και μετά ακολουθούν οι ασκήσεις. Ε, να ρωτήσω συγκεκριμένα, πού ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά αυτό που ρώτησα. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, Αυτά που είπατε και οι δυο σας ε, τα βρίσκω πάρα πολύ καλά και θετικά, αλλά αυτά που μας είπατε στην αρχή, ε, ότι η απειλή μπορεί να είναι και μια φυσική καταστροφή, μπορεί να είναι επιδημίες, φυσικές καταστροφές, αλλά μπορεί να είναι και ανθρωπογενείς απειλές, δηλαδή τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτή νομίζω είναι η σωστή ιεράρχηση. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξής. η απειλές οι οποίες ε, λαμβάνουν χώρα, πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται. Εγώ πρέπει να σας πω ότι για αρκετά χρόνια, ε, μεταξύ άλλων έχω πάει και στο Αφγανιστάν και θυμάμαι ότι το πρόβλημα σε αυτές τις αποστολές ήταν ότι η, λόγω των απειλών τα στρατιωτικά και τα μη στρατιωτικά μέσα ήταν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, είχαμε και το τέταρτο επίπεδο απειλής και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω Αυτή η ροή πληροφοριών ανάμεσα σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δομές, ποια ακριβώ μορφή έχει. Υπάρχει η απαραίτητη τεχνολογία, υπάρχουν ε, μέτρα εξουδετέρωσης γιατί βεβαίως και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν τις δικές τους δυνατότητες ε, αντίδρασης. Και τι γίνεται με τις ε, μη στρατιωτικέ δομές. Παραδείγματος χάρη στην Πολωνία συμβαίνει το εξής. Έχουμε ε, μεραρχίες ή όχι μεραρχίες, με συγχωρείτε, τάγματα και συντάγματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, απειλές. Εγώ θέλω να το πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις απειλές. Το Χαβιέ Νάρτ, είναι άκρος ανησυχητικό. Ε, όλα αυτά που ακούσαμε, που είναι ολόσωστα, αντιστοιχούν, ε, αντιστοιχούν σε κάτι με άλλο που ακούσαμε ότι θα συντονιστούμε, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, ότι θα πρέπει να εξορθολογήσουμε, να ενιοποιήσουμε, να ρέει η πληροφορία. Δηλαδή τι, απέναντι στο τεράστιο πρόβλημα, εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε, ενώ οι άλλοι κάτι κάνουν ήδη. Τι θα πρέπει να κάνουμε μέχρι να είμαστε σε θέση να κάνουμε από τα ιδανικά που μας προτείνεται και τα μέσα στην άμεση πραγματικότητα, γιατί το πρόβλημα το έχουμε χτες, όχι αύριο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η σημαντική σύγκρουση που αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι ένας παραδοσιακός πάνω-κάτω πόλεμος με ένα παραδοσιακό πάνω-κάτω εχθρό. Ο πόλεμος θα είναι με τρομοκράτες ή με αποστολές τα θεραπευτικούς παράγοντες σε ευάλωτες περιοχές όπως είναι η Βόρεια Αφρική. Γι' αυτό ε, δεν βλέπω πραγματική απάντηση απέναντι σε ένα πρόβλημα ε, το οποίο ε, είμαι σίγουρος ότι έχουν εντοπίσει οι τεχνικοί εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια και οι ειδικοί, τουλάχιστον 15 χρόνια. Το δεύτερο αφορά ακριβώς εμάς τους ίδιους και άμεσα και πάλι είναι το τι θα κάνουμε ή το τι κάνουμε ή τι μπορούμε να είμαστε σε θέση σήμερα να κάνουμε. Πολύ καλό είναι ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις χημικές, βιολογικές και λοιπά χημικές ε, πυρηνικές απειλές. Οι πρώτοι όμως που πούλησαν τέτοια τεχνολογία, βακτηριολογική, χημική, ήμασταν οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Οι Ιρακινοί έριχναν χημικά και βομβάρδιζαν από προϊόντα που είχαν πάει από την Ευρώπη και από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία εκεί. Και οι ε, πύραυλοι και οι, οι κεφαλές και οι, θραυσματο... Ε, οι χειροβοβίδες τραυσματοποίησης που χρησιμοποιούσαν ήταν ευρωπαϊκή τεχνολογία. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε τεχνολογία και αυτή πέφτει σε άχαρα χέρια ή σε μη επιδέξια και στο Ιράκ χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται απεμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι ένα υλικό ε, υψηλής διείσδυσης ε, στα ε, άρματα και στα θεθωρακισμένα του εχθρού. Όταν όμως εξαφανιστεί ο εχθρός, παραμένει το απεμπλουτισμένο ουράνιο και μολύνει το έδαφος. Και ο εχθρός εκεί είναι η Δύση θα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον ε, αυτό το εξαιρετικά διεισδυτικό υλικό ή θα σεβαστούμε τη δική μας μεταφυσική ε, στη Δύση. I haven't seen any other indications for uh, colleagues who want to take the floor. Um, I will... Λοιπόν, ε, θα παρέμβω και εγώ και θα ήθελα να πω το εξής ότι <laughs> η γενέτειρά μου είναι το Σόλσμπερι που έχει γίνει και διάσημη πρόσφατα. Ε, εμείς είχαμε να κάνουμε με μια τέτοια επίθεση και πράγματι ήταν ένα από τα ε, πράγματα που κατά την άποψή μου αξίζει να εξετάσει κανείς. Αυτό που εξετάζουμε επίσης είναι η συνεργασία ανάμεσα σε στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αρχές ε, ως απάντηση σε μια τέτοια επίθεση. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε τι μπορεί κανείς ε, να μάθει από ένα τέτοιο γεγονός και όπως είπε και ο συνάδελφός μου ο κύριος Ζέμκε, πράγματι μερικές φορές ε, είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι το Ινστιτούτο του Σόρσμπερι τα, τα έκανε όλα πολύ καλά, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, περιπλοκές ακόμα και μέσα σε ένα κράτος, μέλο. μέλος. Άρα δηλαδή το να συντονίσει κανείς και σε υπερεθνικό επίπεδο ε, τις ε, ενωσιακές δομές, νομίζω ότι αυτό σίγουρα προκαλεί πάρα πολλές δυσκολίες και νομίζω ότι από αυτού πρέπει να βρούμε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εν είδη μιας πρώτης ε, απάντησης, γιατί θεωρώ ότι είναι και πολλοί συμμετέχοντες που και για τις χώρες ε, που τους ενδιαφέρουν μπορούν να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Για τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή, ιδίως ε, διασυνοριακά, Ιδίω εκεί ίσως να υπάρχουν ε, περισσότερα κίνδυνη κίνδυνοι. Κίνδυνοι που συνδέονται ε, με την ε, πυρηνική ενέργεια, με τη χημική βιομηχανία, για παράδειγμα. Πράγματι υπάρχουν, υπάρχει επικοινωνία και διασύνδεση μεταξύ των αρχών και διοικητικών και επιχειρησιακών αρχών, αλλά και ε, υπηρεσιών ε, διάσωσης για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο καθένας. Όταν πρόκειται για άσκηση, για παράδειγμα, στα σύνορά μας, ε, που έχει να κάνει με έναν τεχνολογικό κίνδυνο, όντως, έχουμε τουλάχιστον μία πληροφορία που δίδεται ε, και δίδεται συνέχεια μετά από πλευράς μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πραγματική ε, εμπλοκή και συμμετοχή για τους ε, εταίρους από τη γειτονική χώρα, για το τι θα κάνουν και το καθεξής. Τώρα, για τα διασυνοριακά, αυτή τη στιγμή πράγματι δεν έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σε περίπτωση ορισμένων ε, φυσικών καταστροφών μπορεί να υπάρχει συνεργασία αρκετά διευρυμένη που υπερβαίνει τα σύνορά μας και τα σύνορα άλλων ε, κρατών μελών. Αλλά για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση εδώ των χημικών, βιολογικών και ροδιολογικών και πυρονικών όπλων, υπάρχει σίγουρα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για να έχουμε πράγματι αυτή την επικοινωνία και την επαφή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, Υπάρχουν ήδη ε, πολλές γνώσεις και προετοιμασία γίνεται ήδη ως προς τον προγραμματισμό και ε, τα σχήματα και τις μονάδες που πρότειναν ε, θελοντικά οι ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, η Δανία και η Ιταλία, ε, δήλωσαν ότι όταν υπάρχουν τέτοιες απειλές μπορούν να διαθέτουν μια μονάδα ανείχνευσης και δειγματοληψίας. Και η Δανία πρότεινε μια μονάδα απομόλυνσης. Δηλαδή υπάρχουν ήδη κάποια μέσα που έχουν δηλώσει οι χώρες ότι διαθέτουν. Υπάρχουν και άλλες χώρες όμως που έχουν ικανότητες και δυνατότητες. Και το πρόβλημα ποιο είναι, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν δηλώσει δυνατότητα και προθυμία τα κράτη να τα διαθέτουν αυτά, ότι θα είναι διαθέσιμα τα μέσα ε, σε περίπτωση που χρειαστούν εκτάκτως, γιατί μπορεί να είναι σε κάποια εξωτερική επιχείρηση ή να θεωρούν οι ίδιες σε χώρες ότι κινδυνεύουν από την απειλή και δεν τα διαθέτουν. Έχουν ε, ανταλλαγεί κάποιες προφορίες μετά από το πρόγραμμα δράσης, το αντίστοιχο που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ήταν ε, και στρατιωτικά και πολιτικά όλα μαζί. Καλό θα ήταν να δούμε αμυγός τα στρατιωτικά μέσα ποια είναι. Επίσης ε, γίνονται κοινέ ασκήσεις και γυμνάσια ε, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αρκετά τακτικά. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αυτές οι ασκήσεις αφορούν κάθε φορά μια συγκεκριμένη απειλή και δεν συμμετέχουν πάντα οι ίδιοι. Θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να ασκούνται οι διάφορες ε, μονάδες ε, πολιτικές και στρατιωτικές των κρατών μελών και όχι σε κάποια επιμέρους χρονική στιγμή για μια συγκεκριμένη απειλή. Θα πρέπει αυτό να γίνεται πιο συστηματικά και πιο μακροπρόθεσμα και να, να συμμετέχουν και τα διάφορα επίπεδα από το πιο κοντινό επιχειρησιακό επιτόπου μέχρι το στρατηγικό σχεδιασμό, οι διάφοροι φορείς. Thank you both very much. Thank <laughs> you. Uh, If you Αν έχετε κάποια σχόλια για να ολοκληρώσουμε το θέμα, παρακαλώ. Για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, ε, θέλω να πω ότι ε, ως προς τις ικανότητες αυτές, θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο ε, τις ρήτρες αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης να τις εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος και να δούμε πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα για την ρήτρα αλληλεγγύης ε, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος μέλος, να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεμβαίνει. Και τι σημαίνει αυτό, και εκεί έχει ρόλο να διαδραματίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τα δύο ερωτήματα που έγιναν προηγουμένως σχετικά με τους ε, κανόνες και τα πρότυπα. Πραγματικά εκεί έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Ανάμεσα στα διάφορα πρότυπα ε, και ως προς το υλικό και μόνο, στρατιωτικό και πολιτικό. Ε, και επίση οι ίδιες αποστολές στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Ας πούμε, αποστολή από μόλυνσης ε, θυμάτων από χημικά. Σε στρατιωτικό περιβάλλον ε, απομολύνονται άνθρωποι που φορούν όλοι τα ίδια ρούχα, τις ίδιες στολές και που προστατεύονται. Και αν κάποια στιγμή υπάρχει δυσκολία στην προστασία, ε, είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία που ακολουθούν. Βγάζουν τα ρούχα τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζουν πώς γίνεται κτλ. Και πάντα ο ίδιος. Ε, ε, οι πολίτες είναι εντυμένοι με πολύ διαφορετικό τρόπο. Επίσης έχουμε και παιδιά. Υπάρχει και ένα παιδιατρικό πρόβλημα που είναι πολύ μικρότερο σε στρατιωτικό περιβάλλον. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι οι στρατιωτικοί ε, εταίροι τα ανακαλύπτουν όλα αυτά ε, όταν προσπαθούμε να τους φέρουμε σε μια κατάσταση φυσικής καταστροφής, πολιτικής ε, φύσεως ή καταστροφής, ανακαλύπτουν τα προβλήματα αυτά γιατί δεν τα ξέρουν στο στρατό. Από την άλλη όμως, Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη έχουν αρχίσει και έχουν προχωρήσει και πολύ και αυτό ανάγεται στην απόπειρα την τρομοκρατική του Τόκιο. Πότε ήταν το 1995 όπου τότε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν μόλις αρχίσει να εργάζονται στον τομέα αυτό και όπου γενικά γίνεται καλή δουλειά και συνεργάζονται καλά οι στρατιωτικοί με τους πολίτες. Αλλά έχετε δίκιο που επιμένετε σε αυτό. σε επίπεδο της προετοιμασίας έχει σημασία, δηλαδή Σήμερα, ευτυχώς, ήταν λίγα τα πραγματικά περιστατικά και συμβάντα. Άρα η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών μέσων χωράνε ακόμα βελτίωση. Και γι' αυτό θα πρέπει οι ειδικοί, εκείνοι που έχουν τις ειδικέ γνώσεις για αυτές τις επιχειρησιακές ε, δράσεις, να συναντώνται και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και ε, είναι πάρα πολύ ε, προνομιακός ο χώρος και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεργάζονται και να δουν πώς θα μπορέσουν να προσαρμόσουν τη δουλειά τους έτσι ώστε να συνεργάζονται καλύτερα στρατιωτικοί με πολίτες από τα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση που έγινε για το άμεσο μέλλον, προφανώς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δίνονται εδώ πολύ γρήγορα να αρχίσει η δουλειά. Και πάρα πολύ γρήγορα να συναντηθούν οι ειδικοί και να αρχίσουν να ε, συντονίζονται. Και στα πλαίσια του προγράμματος και της ομάδας που εργάζεται ε, για τα χημικά, βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά όπλα. Αυτή η συμβουλευτική ομάδα που λέγεται Advisory Group για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. να τυποποιηθεί και να εξομαλυνθεί αυτή η δραστηριότητα και να θεσμοθετηθεί το συντομότερο. Με απλό τρόπο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για να μην ε, ε, γενικολογώ. Έχουμε κάποιους που έχουν ε, μολυνθεί από κάποιο χημικό παράγοντα, σαρίν ή υπερίτη. Ορισμένες χώρες προτιμούν να κάνουν την απομόλυνση με πολύ βαρύ τρόπο, με άλλα χημικά προϊόντα. Ενώ άλλα κράτη το κάνουν με πολύ πιο απλό τρόπο, όχι τόσο βαρύ και ε, λιγότερο αποτελεσματικό, αλλά πάρα πολύ γρήγορο. Η αντίδραση δεν είναι ίδια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε σε ένα τέτοιο φόρουμ όπου θα συζητούν αυτοί οι ειδικοί να καταλήξουμε σε ένα κοινό δρόμο που να μην είναι πάρα πολύ περίπλοκος αλλά και εξεζητημένος αλλά μια χώρα που έρχεται να βοηθήσει μια άλλη χώρα να ξέρει τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό η χώρα, τι έκανε τις πρώτες ώρες και τι έχει να κάνει η ομάδα που έρχεται από την άλλη χώρα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, να είμαστε απλοί στην προσέγγιση μας. Thank you. And thank... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο μιλητές για τις ε, εισηγήσεις σας, για το ότι μας ε, παρουσιάσατε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά ευχαριστούμε πολύ και που μας κάνατε και συγκεκριμένες ε, προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό τον τόσο κρίσιμο και περίπλοκο τομέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα κοντά μας. So we will just reorganize the top table, so to speak, and if you can νομίζω ίσως για, κάνα, για λίγο θα κάνουμε ένα μικρό... Thank you. Thank you very much. Right, colleagues. Ε, λοιπόν, συνάδελφοι, δεύτερο τμήμα τώρα της ε, συνεδρίασή μας για σήμερα το απόγευμα με εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την ειδική έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αριστείας στον τομέα των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ε, όπλων. Και ε, συνεχίζουμε την προηγούμενη συζήτηση ουσιαστικά. Με μεγάλη μας χαρά ε, υποδεχόμαστε σήμερα την Πετίνα Γιάκοψεν, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου, που δημοσίευσε πρόσφατα αυτή την έκθεση. Και έχει έρθει ήδη μια φορά φέτος στην συνεδρίασή μας και μας παρουσίασε τα πορίσματα δύο ε, εκθέσεων για τις αποστολές ε, στην περιοχή του Σαχέλ στο Νίγηρα και στο Μαλί. Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε αυτή την έκθεση γιατί συνδέεται και με, τα, με τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένω. παρότι εκεί σταθήκαμε περισσότερο στη στρατιωτική πτυχή της ε, απόκριση, ενώ το ελεγκτικό συνέδριο επικεντρώθηκε στα κέντρα αριστείας που είναι ε, το μεγαλύτερο εξωτερικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι πραγματικά έχουν εντυπωσιαστεί από το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε αυτό το τομέα. Περιμένω λοιπόν με ανυπομονησία να ακούσω την εισήγησή σας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, <laughs> κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτή την ειδική έκθεση ε, για τα κέντρα CBRNN και για τα ε, κέντρα αριστείας. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα βασικό ε, σχέδιο που έχουμε για τους κινδύνους που υπάρχουν και μπορούν να προκύψουν από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Αυτή την πρωτοβουλία την χειρίζεται η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και για την περίοδο 9 ε, έως 19, ε, 13 είχαμε ένα πρόγραμμα τάξης 109 εκατομμυρίων και για την περίοδο 2014-2020 130 εκατομμύρια βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να ισχυθεί η ικανότητα εκείνων των φορέων που ε, είναι αρμόδιοι για να αντιμετωπίσουν χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές και επίση να εστιάσουν και να βελτιώσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές. Ο στόχος ήταν διτός πρώτον να παρακολουθήσουμε τις δράσεις ε, που ε, έχουν αναλάβει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τις συστάσεις από την προηγούμενη έκθεση του 2014. Δεύτερον, να αξιολογηθεί κατά πόσον η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην άμπλυνση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και, και πυρηνικών ε, κινδύνων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα εξετάσαμε, και θα το δείτε αυτό στις διαφάνειες, εξετάσαμε το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν σωστή ε, διαχείριση, στάση διαχείρισης κινδύνου, κατά πόσον η πρωτοβουλία έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε χώρες εταίρου και κατά πόσον υπάρχει και ένα καλό σύστημα αξιολόγηση και ελέγχου για να εντοπίζεται, να αξιολογείται και για να γίνεται και αναφορά σε αυτά τα κέντρα αριστεία σχετικά με τι ε, πρωτοβουλίε. Τι βρήκαμε λοιπόν στην ειδική μας έκθεση. Καταλήξαμε στο ότι η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στο να αμβλύνει πράγματι τους, ε, τις απειλές ε, με τα όπλα CBRN, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν και πολλοί άλλοι κίνδυνοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές έχουν ε, εφαρμόσει τις Κάποιες από τις εκθέσεις ε, που ε, καταθέσαμε έχουν εφαρμόσει μερικά δύο. Ε, τα, οι εταίροι μας ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την εφαρμογή των προγραμμάτων σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό. Υπάρχει ενίσχυση της συνεργασίας και υπάρχει και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Όμως παρά τις προηγούμενες συστάσεις μας για την ιεράρχηση των πόρων στους τομείς που παίζουν ρόλο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει μία ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να κάνει επιλογές με βάση τους κινδύνους. Οι επιλογές δεν γίνονται ούτε με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό ούτε με βάση συγκεκριμένα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στις χώρες εταίρους τα εργαλεία και τη μεθοδολογία για να μπορούν να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να αναπτύξουν ετικά προγράμματα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν κινδύνους από όπλα μαζικής καταστροφής. Βεβαίως η καθοδήγηση για το πώς πρέπει να εντοπίζονται αυτοί οι κίνδυνοι και να ερχούνται δεν είναι ικανοποιητική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ανταποκριθεί αρκετά γρήγορα σε όλους όσοι ζητάνε τη βοήθειά της. Ε, τον Οκτώβριο του 2016, του 2017, ολοκληρώθηκε ο έλεγχός μας. Τέσσερις από 17 χώρες εταίρους είχαν ε, συμπληρώσει το ρητηματολόγιο και μόνο το 31% εξ αυτών είχε καταρτήσει εθνικό πρόγραμμα δράσης. Επίσης διαπιστώσαμε ότι η διαχείριση των πρωτοβουλειών είχε βελτιωθεί. Είχε βελτιωθεί επίσης και η περιφερειακή συνεργασία. Παραμένουν όμως ακόμα σημαντικά εμπόδια. Η πρωτοβουλία αυτή έχει βελτιώσει ε, τη συνεργασία, αλλά ε, πάρα πολλές αρχές ε, είναι χρονοβόρες και χρειάζεται αρκετό καιρό για να εφαρμόσουν τα προγράμματα. Εξαιρουμένης μίας, όλες οι άλλες δεν έχουν ένα κομβικό, ένα κέντρο για να μπορούν να διασφαλίσουν τη συνεργασία. Τα προγράμματα έχουν αποδώσει και οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις ασκήσεις βελτίωσης της ικανότητας. Όμως, τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν είναι προτεραιότητα σε χώρες που συνεργαζόμαστε. Ε, τα ε, κομβικά, τα κέντρα μάλλον, τα εθνικά που θα πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο στα όπλα μαζικής καταστροφής δεν ε, δίνουν την απαραίτητη εξοδότηση στα κράτη-μέλη. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική βούληση. Και από τότε που πρωτοκαταθέσαμε τις ειδικές μας εκθέσεις, οι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν περισσότερο, αλλά διαπιστώσαμε ότι δεν είναι ικανοποιητικά ενεργές για να προάγουν τις πρωτοβουλίες και τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν περιλαμβάνουν συστηματικά στην πολιτική, την ασφάλεια ή τον πολιτικό διάλογο. Τα εθνικά προγράμματα δράσης αναφέρουν πολλές δράσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από εθνικούς προϋπολογισμούς. Παρόλα αυτά διαπιστώσαμε ότι οι συνέργειες δεν την χάνουν πλήρης εκμετάλλευσης και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις Γενικές Διευθύνσεις Επιτροπής και στους δωρητές είναι περιορισμένη. Ε, κυρίως ε, ε, περιορίζονται όλοι στα υπάρχοντα κονδύλια. Ένα βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η περιφερειακή συνεργασία. Τα εθνικά κέντρα συναντιόνται για να συζητήσουν κοινά σημεία και απόψεις για προγράμματα. Η πρόσφατη ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων σε περιφερειακό επίπεδο αποδείχθηκε πάρα πολύ ε, χρήσιμη. Παρόλα αυτά, οι χώρες εταίροι που επιθυμούν ε, να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, θέλουν να αντιμετωπίσουν πρώτα τις δικές τους ανάγκες. Ως εκ τούτου, περισσότερες δραστηριότητες παραμένουν σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχει περιφερειακή συνεργασία. Άρα, δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες περιφερειακές συνταλλαγές και βέλτιστες πρακτικές. Εξάλλου, υπάρχει και η ανάγκη να ε, καθορίζεται ποιος και να καθοδηγείται η πολιτική, ε, να υπάρχει σαφέστερος ε, έλεγχος, γιατί δεν είναι ικανοποιητικό ο έλεγχος, ούτε η αξιολόγηση. Η τεκμηρίωση δεν είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι, ούτε δείκτες, ούτε και σωστή συγκέντρωση δεδομένων. Έτσι λοιπόν καθίσατε πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις μιας πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου δεν είναι ακόμα δυνατόν να αξιολογηθούν οι πόροι για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν βελτιωθεί οι ικανότητες για να αμβληνθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα όπλα μαζικής καταστροφής. Τι προτείνουμε λοιπόν στην ειδική μας έκθεση. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την πρωτοβουλία και συστήνουμε η Υπηρεσία εξωτερική δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να ε, ε, κάνουν την ιεράρχηση ε, με βάση την αξιολόγηση, να ενισχύσουν την περιφερειακή διάσταση, να ενισχύσουν περαιτέρω το ρόλο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβουλία, να εντοπίσουν κάποιες συνέργειες και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία, να είναι ορατές οι πρωτοβουλίε και τέλος, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει το, η πύλη αυτή ε, της πρωτοβουλίας που θα επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε όλες ε, τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχουν δεχθεί όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και με πολύ μεγάλη μου χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας για αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσταν ιδιαίτερα σαφείς στην παρουσίασή σας, αλλά και η ίδια η έκθεση. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Θα μιλήσω γερμανικά αυτή τη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εντύπωσή μου λοιπόν είναι ότι ε, η τελική σας, το τελικό σας πέρασμα είναι καταστροφικό όσον αφορά το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής ε, προστιθέμενης αξίας. Εσείς είπατε ότι ε, το θέμα αυτό δεν έχει καμία προτεραιότητα. Επίσης, είπατε ότι ούτε καν μπορούσατε να διαπιστώσετε ορισμένα πράγματα, ούτε καν μπορέσατε να διαπιστώσετε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Διερωτώ με λοιπόν, γιατί πραγματικά νιώθω κάποια μηχανία. Διερωτώ με πώς ε, μπορεί κανείς να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη, να προκαλέσει κανείς το ενδιαφέρον τους, έτσι ώστε μέσα από πιο στενή συνεργασία και με το να αποδώσουν περισσότερη προσοχή σε όλα αυτά τα προγράμματα ή στην πρωτοβουλία, πώ είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να προκύψει θέμενη αξία. Βεβαίω και δεν μπορεί κανεί να το εξαναγκάσει ενδεχομένω το θέμα αυτό για πάρα πολλά κράτη-μέλη να εξακολουθεί να είναι πολύ αφηρημένο γιατί αν κάποιος ο ίδιος δεν έχει εκτεθεί ε, σε μία επίθεση τότε την κλίμακα των προτεραιοτήτων του, το θέμα αυτό πάει πολύ χαμηλά. Πραγματικά μου προκαλέσατε μηχανία. Ναι, μεν μας παρουσιάσετε όλες αυτές τις πολύ ωραίες συστάσεις, αλλά τώρα κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα τις λάβουν υπόψη τους. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εσείς ε, βεβαίως απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κατ' ουσίαν ε, τελικά πρέπει να δραστηριοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Και αν δεν το κάνουν, τι να κάνουν και οι Με λύπη μου το διαπιστώνω αυτό, αλλά ε, ίσως και να μην τα κατάλαβα καλά, και να μου τα πείτε τώρα εσείς καλύτερα, να τα καταλάβω καλύτερα, αλλά φοβάμαι ότι ε, μάλλον δεν πρέπει να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Για να δω. Μάικλ, νομίζω ότι μόνο εσύ ήθελες να πάρεις το λόγο. Και εγώ βέβαια, αναπόφευκτα θα πάρω το λόγο. Έχετε εντοπίσει ξεκάθαρες ελλείψεις σε ό,τι αφορά την σημερινή μας λειτουργία και αντιμετώπιση και κατά τη γνώμη μου τίθεται και ζήτημα ιδιοκτησίας. Ποιος θα αναλάβει και θα ενστερνιστεί αυτή την ευθύνη και αρμοδιότητα. Ναι, βέβαια, με καλύτερη καθοδήγηση και το καθεξή. Αν πρέπει να είναι περισσότερο ζήτημα αντιπροσωπιών, ε, περισσότερο θέμα της Γενικής Διεύθυνσης, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο υφιστάμενο πρότυπο ή μοντέλο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο, το οποίο όμως να μπορεί να εφαρμοστεί και στα κέντρα αριστείας. Ένα θετικό παράδειγμα λοιπόν προς μίμηση, που να πούμε να ορίστε, αυτό λειτουργεί, ας το εφαρμόσουμε και εδώ. Δεν ξέρω, έτσι το ρωτάω. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Ένα από τα βασικά απορίσματα ε, τη έκθεση είναι ότι πράγματι υπάρχει περιθώριο βελτίωση και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πλευρά αντιπροσωπιών. Γιατί υπάρχουν υψηλέ προσδοκίε από τι χώρε εταίρους μα και θα ήθελαν πραγματικά να συμμετάσχουν, αλλά ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι να ε, εξεταστεί κάθε αίτηση και να αρχίσει το κάθε project. Και ίσως ε, θα ήταν καλύτερο να αντλήσουμε ένα από διδάγματα από τις ε, εμπειρίες του άλλου. Αλλά μας παίρνει περίπου δύο χρόνια για να μπούμε σε αυτόν τον κύκλο άντλησης διδαγμάτων από τα project έχουμε δει ότι έχει δημιουργηθεί όμως μια κουλτούρα ασφάλειας και προστασίας. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική και εμείς στις συστάσεις μας ε, λέμε ότι θα πρέπει να βασιστούμε πάνω σε αυτή τη δυναμική. Ότι οι χώρες εταίροι πραγματικά ακτιμούν τα όσα έχουν γίνει, αλλά και να επιταχύνουμε λίγο τη διαδικασία, να μάθουμε ένας από τον άλλον και από τις εμπειρίες μας γιατί τα όσα μας μεταφέρονται από τις χώρες εταίρους ως θετικά σημεία είναι οι επιχειρήσεις αύξησης ικανοτήτων. Και όταν έχουμε αυτές τις ε, κοινέ ασκήσεις, βλέπουμε ότι οι συμμετέχοντες ε, ασχολούνται πολύ περισσότερο και μεταφέρουν τα όσα έχουν γίνει εκεί και πιέζουν να επαναληφθεί το ίδιο σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, είναι περιορισμένοι πόροι και έτσι μπορεί να είναι δύσκολο να πετύχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για όλες τις χώρες εταίρου ταυτόχρονα. Γιατί δεν έχουμε παρκεί πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Μιλήσατε, Πρόεδρε, για την ε, εφαρμογή θετικών εμπειριών ε, εδώ. Πράγματι, βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες θετικές εμπειρίες σε κάποια project και βλέπουμε ότι για κάποια project, επειδή δεν υπήρχε σωστή τεκμηρίωση ε, στην διαδικτυακή πύλη, ε, ξαναέγινε, επανελήφθηκε η διαδικασία. Αντί δηλαδή να μάθουμε κάτι από την προηγούμενη εμπειρία, υπήρξε μια τέτοια σπατάλη χρημάτων γιατί πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή. Επομένως υπάρχουν τέτοια θετικά ε, παραδείγματα και μοντέλα και πρέπει αυτά να μπορούν να επαναληφθούν. Πρέπει η πύλη να βελτιωθεί πολύ για να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των εταίρων στην πληροφορία, γιατί αυτό είναι βασικό στοιχείο της όλης αυτής της διαδικασίας. Ελπίζω έτσι να απαντώ στο ερώτημά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι. Ευχαριστούμε πολύ, πράγματι. Είστε τόσο αποτελεσματικοί και σαφείς στις απαντήσεις σας, που θα σας αφήσουμε να φύγετε και λίγο πιο νωρίς. Εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε. Can I Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Γιάκοψεν.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 Right, colleagues. Uh, Ωραία, συνάδελφοι. Ας περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος ε, της συνεδρίασής μας για σήμερα το απόγευμα. Αφήνουμε κατά μέρος ε, τα προηγούμενα θέματα. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ιούχαν Πάρτς, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. και είναι αρμόδιος για την ε, πρόσφατη έκθεση για την Αφρικανική Αρχιτεκτονική ε, Ασφάλειας Ειρήνης και Ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντική γιατί αύριο θα εξετάσουμε ε, τον μηχανισμό ειρήνης που θα συμπεριλαμβάνει και το συγκεκριμένο Γι' αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερω. Για τη δεύτερη πρόταση, συμφωνείτε μαζί μου, φαντάζομαι, ότι ο προβλεπόμενο ρόλο του Ελληνικού Συνεδρίου για το μηχανισμό λογικά θα συνάδει πλήρω και με τη διαδικασία απαλλαγή ε, και του ρόλου απαλλαγή, μάλλον που δίνει το Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή όμω δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση. Και πάλι με τα χαράς βλέπουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, διενεργεί αυτούς τους ελέγχους σε έναν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και εκτιμούμε και τη βούλησή σας να είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να τα συζητήσουμε. Σε εμά βέβαια η ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι αυτή που διδαμετίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Παρακολουθείτε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Καταλαβαίνω ότι για σας δεν είναι εύκολο να περνάτε από το ένα σημαντικό θέμα στο άλλο, αλλά επιτρέψτε μου ε, να μιλήσω με λιγότερο τεχνικούς ε, όρους για να συνεννοηθούμε περισσότερο. Πρώτον, το ελεγκτικό συνέδριο έχει θέσει μια σειρά προτεραιότητες. Για χρόνια, μία από αυτές τις προτεραιότητες είναι η στόχευση στον τομέα της ασφάλειας, από όπου προκύπτουν και πολλοί, πολλές απειλές και κίνδυνοι. Είχαμε και εξελίξεις στην Αφρική και σίγουρα θα έχετε δει και μία σειρά εκθέσεις για διάφορες πτυχές ε, παρέμβασης ε, της Ευρώπης ε, στην Αφρική, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίω ό,τι αφορά τη διευθέτηση για την ασφάλεια στην Αφρική, που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο είχατε δυνατότητα να τη διαβάσετε. Έχουμε και μικρότερες... Προσπαθούμε να έχουμε σύντομα κείμενα και πιο εύληπτα. Το ένα ζήτημα αφορά την ε, απόδοση. Πώς η μακροπρόθεσμη ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θέσπιση αυτού του αρχιτεκτονήματος ε, στην Αφρική, πώς ακριβώς επιτυγχάνει τα αποτελέσματα και τους στόχους που έχουν διακηρυχθεί πολλές φορές εδώ και πολλά χρόνια. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με το ζήτημα της ε, ε, χρηματοδότησης. Εγώ θα σταθώ στο πρώτο όμως. Και θα σας παρουσιάσω τα συμπεράσματά μας. Είναι λοιπόν δύο τομείς που σαφώς ε, και είναι αλληλένδετοι, αλλά πιστεύω ότι και εσείς ως μέλη του Κοινοβουλίου που ασχολείστε συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας σας ενδιαφέρουν περισσότερο. τα συζητήσαμε και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. Και είχαμε και μία συνάντηση στην ε, Παναφρικανική Ομάδα του Κοινοβουλίου και εκεί συζητήσαμε και αυτή την έκθεση. Αυτά είναι η εισαγωγή. Το βασικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή στήριξη προς το αφρικανικό αρχιτεκτόνημα ειρήνη και ασφάλεια είναι ότι πρόκειται για μία ε, συγκέντρωση δυνάμεων. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές και με την υπηρεσία εξωτερική δράση και είμαι βέβαιο ότι ε, δεν ε, τους ικανοποιούν τα πράγματα και η βασική μας σύσταση θα το πω και στη συνέχεια βέβαια, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική παρέμβαση στην, ε, στο αφρικανικό αρχιτεκτόνημα θα πρέπει να επανεξεταστεί. Δεν θέλουμε βέβαια να αναλάβουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως είναι σαφές ότι αυτή η στρατηγική που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια ή και με άλλους ε, δωρητές, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει το επιχειρησιακό κόστος του προσωπικού και ούτε καθεξής τεχνικών θεμάτων, δεν λειτουργεί. Εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην δημιουργία δυναμικού, είτε σε επίπεδο Αφρικανικής Υπήρου, είτε σε περιφερειακό, είτε και στο τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το βασικό μας πόρισμα. Τώρα για το πλαίσιο της ΑΠΣΑ. Έθεσε εξ αρχή το 2002, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν ε, είχε εμπλακεί ε, στο μηχανισμό άψα, είναι ότι ήταν ένα εργαλείο με βασικό στόχο οι ίδιες οι αφρικανικές χώρες να έχουν τις δυνατότητες, την ικανότητα να αποτρέπουν και εάν αυτό είναι απαραίτητο, να ενεργούν για τη διασφάλιση της ε, ειρήνης και ασφάλειας στην Αφρική. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το μέγεθος της Επίρου και τις εξελίξεις εκεί. Και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούν να μας δείξουν κατά πόσο και πότε μπορούμε να αξιοποιούμε το αφρικανικό αρχιτεκτόνομα. Νομίζω λοιπόν ότι μία από τις βασικές προκλήσεις είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι δημιουργούνται μικρές δομές σε μια τεράστια ήπειρο, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή προβλημάτων, αλλά και την ε, διασφάλιση της ασφάλειας σε όλη την Ήπειρο. Το πιο σημαντικό λοιπόν αίτημα είναι αυτό που πλευράζει δωρητών προς τους Αφρικανούς. Παρουσιάζουμε και μια επισκόπηση των εξελίξεων και της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Ε, τα πράγματα επιδεινώνονται αυτή τη στιγμή. Αν δούμε λοιπόν τον αριθμό των ε, συγκρούσεων, πολέμων και ούτω καθεξής με βάση της διεθνούς ε, κλίμακας και βαρομέτρου, έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις. Από 67 πήγαμε στους 73 σε σχέση με το 16-17. Και έχουν αυξηθεί και οι μικρής κλίμακα πόλεμοι. Από 7 έχουν πάει στους 10. Παρά τις προσπάθειες των δωρητών και άλλων εταίρων, βλέπουμε ότι δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των κρίσεων είναι ακόμα αυξητική η τάση. Πρέπει μετά να κατανοήσουμε σαφώς τις αιτίες των συγκρούσεων. Δεν πρόκειται για κάτι καινοφανές. Ε, πρέπει να αξιολογήσουμε παρκώς τις στρατηγικές ε, των δωρητών και να τις λάβουμε υπόψη τρεις βασικές αιτίες. Ε, μεταβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων, ε, διακρατικές συγκρούσεις και εξωτερικές επιρροές. Είναι οι τρεις βασικές αιτίες συγκρούσεων. Αλλά έχουμε και την μητέρα όλων των αιτιών. Που είναι οι αδυναμίες των κρατών. Μία από τις βασικές αιτίες ε, αστάθεια στην Αφρική. Γιατί συχνά έχουμε διεφθαρμένες ε, κυβερνήσεις που οδηγούν και σε αδύναμους ε, μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί βασικός ε, φορέας λήψης αποφάσεων στην Αφρικανική Ήπειρο, το Συμβούλιο Ασφάλειας και Προστασίας, ε, Ειρήνης και Ασφάλειας, εκπροσωπεί χώρες που έχουν ε, καταρρύψει, δεν ε, τηρούν ε, τις ίδιες τις αρχές που έχουν θεσπιστεί. Πρέπει λοιπόν αυτό να το έχουμε κατά νου. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εστιασμένη προσέγγιση για την προσφορά λύσεων. Δυστυχώς, η έκθεσή μας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τη προσπάθειες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Επιτροπής Εξωτερική Δράση, ότι πρέπει να υπάρχει σαφέ σημείο εστίαση, χάραξη και θέσπιση προτεραιοτήτων που είναι δύσκολο να τα συμφωνήσουμε με όλα αυτά. Μετά δεν υπάρχει συνέπεια στις αποφάσεις για το κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθούν νέες ικανότητες σε ε, υπηρετικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί σε, μη, σε έναν κατακαιρματισμό και ε, διασπορά των ε, προσπαθειών και έτσι δεν πετυχαίνουμε αυτά αποτελέσματα. Βασικές τώρα παρατηρήσεις και πορίσματα ως προς τον άψα σε ό,τι φορά αρχικά την ιδιοκτησία του αφρικανικού αρχιτεκτονήματος. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Το 2002, όταν δημιουργήθηκε το Αφρικανικό Αρχιτεκτόνημα, είχαμε μία σειρά ερευνών, ελέγχων που, δεν, που έλεγαν ότι δεν αναλάμβανε κανείς ε, την ιδιοκτησία του άψα και έτσι δεν ήταν βιώσιμος ο μηχανισμός. Υπήρχαν ε, προσπάθειες γιατί αν είχαν φύγει κάποιοι φορείς θα είχε καταρρεύσει όλη η προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε να, αν σταματούσε να χρηματοδοτεί κάποιες δομές απλά θα κατέρεαν ιδίως σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Φυσικά, βασικός ιδιοκτήτης του προγράμματος πρέπει να είναι τα κράτη της Αφρικής, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτή την ε, συνεισφορά και συμβολή θα πρέπει να ε, έχουμε κατά νου κατά πόσο προάγεται η εθνικο επιπεδο φυσικα βασικος ιδιοκτητη του προγραμματος πρεπει να ειναι τα κρατη της αφρικης αλλα δυστυχω αυτο δεν ισχυει βλεπουμε λοιπον οτι με αυτη την συνεισφορα και συμβολη θα πρεπει να εχουμε κατα νου κατα ποσο προαγεται η ιδιοκτησια των Αφρικανικών κρατών ε, ως προς τον άψα. Την τελευταία πενταετία όμως βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πόροι βασίζουν τεχνικά κόστη, ε, βασική συνεργασία και ούτω καθεξής. Επομένως, μειώνεται, δεν αυξάνεται η αφρικανική ιδιοκτησία του προγράμματος. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει επανεστίαση στις, στην αύξηση ικανοτήτων και να ζητήσουμε ή να απαιτήσουμε από τα αφρικανικά κράτη να αναλάβουν μεγαλύτερο κομμάτι του κόστους και της ιδιοκτησίας ε, του προγράμματος. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο μέλλον για την οικοδόμηση δυναμικού και για την ε, ασφάλεια. Το αφρικανικό αρχιτεκτόνημα έχει μία σειρά στοιχεία και στην έκθεση θα βρείτε βέβαια πολύ περισσότερα στοιχεία για την σημερινή κατάσταση. Να έχετε κατά νου ότι αυτά είναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα ε, εξελίξεων δεκαετίας. Σε ό,τι αφορά την ε, απρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων, έχουμε μία σειρά ε, προσεγγίσεις. Αρχικά έχουμε μόνο ένα άτομο που ασχολείται με τη διαμεσολάβηση, την πρόληψη κ.ο.κ. Για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, από τεχνικής άποψης λειτουργούν, αλλά υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στην αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχει σημαντικό κενό μεταξύ τη έγκαιρη προειδοποίηση και έγκαιρη απόκριση, γιατί δεν υπάρχουν αρκετέ συνδέσει μεταξύ ε, των εθνικών και ευρύτερων ε, συστημάτων έγκαιρη προειδοποίηση. Και μετά υπάρχει και ένα άλλο κενό ε, σε ό,τι αφορά την χρήση των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν συλλεγεί. Τρίτο στοιχείο είναι η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και το σχετικό τμήμα ειρήνης και ασφάλειας. Είναι μια βασική δομή με μια σειρά ρόλους σε ό,τι διαχείριση και συντονισμό, αλλά υποχρηματοδοτείται από την Αφρικανική Ένωση. Το 2010 οι δωρητές αποφάσισαν να σταματήσουν να καλύπτουν ε, τα βασικά πιασιακά κόστη, όμως Υπάρχουν ε, σημαντικές ελλείψεις σε άλλους κλάδους και είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να τα δείτε ε, όλα αυτά στην έκθεσή μας. Αναλύσαμε ποιοι είναι αυτοί που εργάζονται σε αυτές τις βασικές ε, δομές. Πρόκειται για ειδικού στον τομέα της ειρήνης και ασφάλειας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλύπτει ε, τους μισθούς τους. Σε ό,τι αφορά την ε, απόκριση του Συμβουλίου Ειρήνης ε, και Ασφάλειας, υπάρχουν διάφορα προβλήματα που το επηρεάζουν υπάρχουν και κάποιοι σκληροπρινικοί, ας πούμε, ηγέτες που εξακολουθούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο και ε, προσποιούνται ότι επιλύουν ζητήματα που άπτονται της ειρήνης, των δικαιωμάτων και της ασφάλειας. Όμως υπάρχει έλλειψη βούλησης σε κάποια κράτη ε, να λάβουν θέση όταν ε, θεωρούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους ή όταν δεν θέλουν να έρθουν σε άμεση αντιπαράθεση με άλλα κράτη. η μονάδα η δύναμη επιφυλακής ε, δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί από την Αφρικανική Ένωση μέχρι τώρα, καθώς ε, το πληροφορικό σύστημα δεν είναι ακόμα επιχειρησιακό ε, και δεν υπάρχει έτσι δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης δυνάμεων εξαιτία υλικοτεχνικών περιορισμών. Τέλος, έχουμε την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη μετά τη σύγκρουση. Βλέπουμε ότι είναι ε, το λιγότερο αναπτυγμένο ε, μέρος της άψα. Στην έκθεσή μας έχουμε επισημάνει και μια σειρά προκλήσεις ε, για το άψα. Θα τα απαριθμίσω εν συντομία. Πρώτον, έχουμε την χρηματοοικονομική και θεσμική ικανότητα των βασικών φορέων της Αφρικανικής Ένωσης και των περιφερειακών οργανώσεων που είναι αδύναμες, πρέπει να ενισχυθούν. Και το βασικό ερώτημα είναι η διασύνδεση μεταξύ τη Αφρικανική Ένωση και αυτών των, Αφρικανικής Ένωσης και αυτών των οργανώσεων. Πολλά θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν ε, για να αποφευθούν οι άλλοι επικαλύψεις ως προς την ε, επικουρικότητα. Υπάρχει λοιπόν πάντα μια σύγχυση για το ποιος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα κάθε φορά. Σε ποιο επίπεδο δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε στην ε, ανάπτυξη ε, ικανοτήτων και τι υπό στρατηγικής άποψης είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Ανέφερα ήδη την έλλειψη πολιτικής βούλησης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε περιπτώσεις κρίσεων και δεν υπάρχει και μηχανισμός επιβολής των αποφάσεων που έχει λάβει το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας. Πριν ολοκληρώσω πρέπει να πω ότι έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους σε διάφορες αφρικανικές χώρες και την Αφρικανική Ένωση συμφωνούν πάρα πολύ με τις παρατηρήσεις μας και τις συστάσεις μας και τα κριτήριά μας. Παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος έλλειψης επικοινωνίας Ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα αποτελέσματα άψα δεν έχουν ε, υλοποιηθεί με τρόπο συστημικό, συστηματικό και υπάρχουν ειδικέ προτεραιότητες. Ε, εμείς λέμε ότι δεν έχετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι βεβαίως και έχουμε. Λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει με τρόπο αποτελεσματικό ε, την Αφρική και η στήριξη του μηχανισμού άψα είναι ένα έργο μακράς πνοής που δεν μπορούν τα αποτελέσματά του να μετρηθούν άμεσα. Υπάρχει μια αναντιστοιχία στις διαπιστώσεις μας. Για μας αυτά τα στοιχεία δεν ε, μπορώ να πω ότι μας εκπλήσουν, αλλά μας ανησυχούν κάπως. Γιατί έχουμε 14 συμβάσεις και θα πρέπει να δούμε πώς αντανακλούν εκεί τις προτεραιότητες άψα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει βεβαίως ότι έχει ε, σαφείς προτεραιότητες. Βρήκαμε ότι σε 8 περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα κονδύλια στον προϋπολογισμό δεν επέτρεπε να δούμε και να διαπιστώσουμε ποια κονδύλια πηγαίνουν σε ποιες προτεραιότητες και πυλώνες άψα. Βεβαίως υπάρχει ένας οδικός χάρτης 2016-2020, έτσι ευρύτατος τα Και, και έχετε συμμετάσχει κι εσείς στην κατάρτισή του. Αλλά έχει πέντε προτεραιότητες και ε, μύριους στόχους και αποτελέσματα, αλλά θεωρείται πάρα πολύ περίπλοκο για να εφαρμόζεται στην πράξη ως εργαλείο και η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης φαίνεται ότι δεν ε, το έχει κάνει ακόμα κτήμα της. Και αυτό δεν είναι δική μας μόνο παρατήρηση, αλλά και μια ε, παρατήρηση ε, που έχει κάνει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από στις στι υπηρεσίε τη. Υπάρχει ο ειδικός χάρτης, χάρτη, καλύπτει πάρα πολλά στοιχεία, αλλά είναι πληθώρα οι στόχοι, οι δράσει, οι δραστηριότητε κτλ. Και χάνεται εκεί η προσπάθεια. Και είναι σημαντικό αυτό στη συνεργασία μας με την Αφρικανική Ένωση. Τρίτον, Έχουμε διαπιστώσει ότι ο έλεγχος μας βασίζεται κυρίως στις δραστηριότητες οι οποίοι αναπτύχθηκαν, μέχρι το 2014, αλλά αναλύσαμε και το ευρύτερο πλαίσιο και έτσι πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι η άψα ξεκίνησε ήδη το 2008, άρα δηλαδή ήδη υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα θα έπρεπε να είναι πιο όρατα επειδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια. Και τέλος, η καταβολή των μισθών και άλλες, ε, λειτουργικά, και άλλες λειτουργικές δαπάνες για μία σειρά αξιωματούχων ε, σίγουρα είναι διαφορετικό όλο αυτό σε σχέση με το παρελθόν, αλλά επίσης θέλω να πω ότι πολύ, πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί εάν υπήρχε η σωστή προσέγγιση και η τήρηση των προϋποθέσεων. Ε, τέλος, δεν θα σας διαβάσω τις συστάσεις μας, αλλά ε, θα ήθελα όσον αφορά τις συστάσεις να υπογραμμίσω τρεις λέξεις. Ρεαλισμός, ιδιοκτησία και βιωσιμότητα. Ο ρεαλισμός πρέπει να είναι η ε, κατευθυντήρια αρχή για να κατανοήσει κανείς τις ικανότητες που, πρέπει, που είναι απαραίτητες ε, και πρέπει να υπάρχουν σε κάθε επίπεδο. Εμείς συστήνουμε να ξεφύγουμε ε, από την υποστήριξη επιχειρησιακών ή λειτουργικών, τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και να περάσουμε σε μέτρα βελτίωσης της ικανότητας. Όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με την διοκτησία του προγράμματος, πρέπει ε, τα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης πρέπει να έχουν το πρόγραμμα αυτό να το οικειοποιηθούν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα με 0,2% ε, τέλος ε, για να χρηματοδοτηθεί ο λειτουργικός προϋπολογισμός και το Ταμείο Ειρήνης, αλλά η εφαρμογή όλων αυτών παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το μέλλον. Εμείς ε, προτείνουμε να ελέγχετε το πρόγραμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες ότι ε, θα έχουμε μία βιώσιμη λύση για τη χρηματοδότηση των ε, βασικών ε, δαπανών των Αφρικανικών κρατών. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί καταδεικνύει τη βούληση, την οικειοποίηση για θέματα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε για αυτές τις ε, ειλικρινείς σας εξηγήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της ε, δουλειάς σας. Θα έλεγα, επειδή ξεκινήσαμε λίγο νωρίς και ήθελε να έρθει, να έρθει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τελικά έρχονται, είναι καθοδόν από ό,τι μας είπαν και θα πούν και εκείνη την άποψή τους. Σε αυτό το σημείο ξέρω ότι ο συνάδελφός μου, ο κύριος Γκάλερ θέλει και αυτός να θίξει ένα θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται. Η Επιτροπή πάντα μπορεί να λέει ότι κάπου εδώ είναι μέσα στην πόλη στις Βρυξέλλες, γιατί εδώ βρίσκονται. Σα ευχαριστούμε πολύ για την εκθεσή σα. Πρέπει να σα πω ότι έχω και κάποιες αφρικανικές ιδιότητε Με την έννοια ότι διάβασα αυτή την εκθέση πριν από τρει εβδομάδες, αυτή την πολύ μεγάλη διάρκεια πτήση μου ε, προς το Johannesburg. Ε, συμμετέχω ε, στην Επιτροπή Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες και σε πολλές άλλες ενώσεις και αυτό το άψα ε, συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες και νομίζω ότι εσείς πολύ σωστά παρουσιάσατε ε, τα αίτια Πολύ σωστά τα είπατε αυτά που είπατε για την Αφρική και γι' αυτό ε, και εγώ τη διάβασα την έκθεση ε, και την ε, μοιράσαμε και στο Ιωάννεσπουργκ σε μία μελέτη που κάναμε για να αναλύσουμε τα αίτια της κρίσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση. Δεν είναι ότι κάνετε απλά μία έκθεση και εμείς τη μοιράσαμε. Ε, μας ενδιαφέρουν και δουλεύουμε πάνω στα συμπεράσματά σας. Εκείνο το οποίο βιώνουμε είναι ότι πράγματι υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός ε, ότι πρέπει να βρεθούν αφρικανικές λύσεις στα αφρικανικά προβλήματα και να υπάρχει ένα τέτοιο αρχιτεκτόνημα, αλλά όταν τα πράγματα γίνονται πιο συγκεκριμένα και όταν προκύπτει κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, τότε συνήθως υπάρχει έλλειψη πόρων, ε, υπάρχει έλλειψη πολλών ε, συστατικών που θα μπορούσαν να καταστήσουν μια επιχείρηση επιτυχημένη. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλά από τα θέματα ε, που θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό, ε, δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν. Παραδείγματο χάρη γίνεται λόγο για μια δύναμη επιφυλακής για την Αφρική. Και υπάρχει επιθυμία να συσταθεί μια τέτοια επιτροπή μια τέτοια δύναμη, απλά δεν υπάρχει όμως. Και ένας από τους λόγους είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ε, και δεν υπάρχει και η δέσμευση να δουλέψει κανείς πάνω σε αυτό. Εάν λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε χρηματοδοτήσει έστω τα βασικά και δεν έχουμε αποκτήσει προστιθέμενη αξία, εμπειρία, αλλά όπως σας λέω ε, υπάρχουν απλά κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι, ε, τότε και από πλευράς Αφρικής δεν μας παίρνουν ε, σοβαρά για να κάνουν και αυτό που εκείνοι εννοούν. Και με την έννοια του να συστήσουν ένα τέτοιο αρχιτεκτόνημα ή μία δύναμη επιφυλακής ή να εξετάσουν επίγοντα θέματα με επιχειρησιακό τρόπο. Κάτι που θα ήταν απαραίτητο. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και όχι μόνο γιατί λέμε στους Αφρικανούς ότι δεν θα ανακατευτούμε πια, αλλά για να τους υπενθυμίσουμε ότι είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τις δικές μας τις ευθύνες. Θα ήθελα λοιπόν η υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερικής, η επιτροπή, υπηρεσία εξωτερικής δράσης να υιοθετήσει τις ε, συστάσεις σας και να καταστήσει σαφές στην Αφρικανική Ένωση ε, το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους. Δεν έχω ακόμα σχηματίσει άποψη για το εξή και αυτό είναι ένα ερώτημα. Αναφερθήκατε και στις ε, υποπεριφερειακές οργανώσεις, έχουμε στο νότο, έχουμε στην ανατολική πλευρά της Αφρικής και έχουμε και ε, κάποιους ε, ad hoc ε, οργανισμούς που και αυτοί αναλαμβάνουν το ρόλο να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν του Ιμπόκο Χαράμ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Ε, θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που συμβαίνει αυτό. Αλλά μερικές φορές διερωτώμε κατά πόσον ίσως θα ήταν πιο σοφό να βασίζεται κανείς σε αυτούς τους υποπεριφερειακούς όπως αποκαλούνται οργανισμοί. Γιατί από τη μια ε, τα κράτη είναι πιο κοντά στο πρόβλημα και στην κρίση και αυτό είναι το θετικό στοιχείο του να λαμβάνει κανείς περισσότερες ευθύνες. Το άλλο είναι ότι αν είναι κάποιος πολύ κοντά σε όλα αυτά, τότε ενδέχεται να έχει και μία δική του κρυφή ατζέντα, ένα κρυφό θεματολόγιο. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα οι Αφρικανοί κατά πόσον τηρουμένων των αναλογιών θα προτιμούσαν να έχουν ομάδες ή συμβουλές που να δοθούν από μακριά ίσως, όχι από τους ίδιους Αφρικανούς ή μήπως προτιμούν να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητε οι πιο κοντινοί τους γείτονες που αυτοί όμως μπορεί να έχουν ε, δική τους ατζέντα. Ε, δηλαδή προτιμούν να υπάρχει περιφερειακή οργάνωση ή παναφρικανική οργάνωση. Αυτά έχουν και υπέρ και κατά. Όταν είναι κανείς πιο μακριά δεν ασκείται πολιτική πίεση εκτός από το γενικότερο αίσθημα των αισθάνονται όλοι ότι ανήκουν στην Αφρική. Ε, σε αυτήν λοιπόν τη φάση βρισκόμαστε. Νομίζω η πραγματιστική προσέγγιση είναι ότι λόγω της κρίσης ε, και όταν λέμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, ε, τότε ενδεχομένως θα πρέπει και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί βεβαίως η εναλλακτική λύση είναι ότι αν δεν βοηθήσουμε τους Αφρικανούς να λύσουν τα προβλήματά τους, τότε προφανώς αυτά τα προβλήματα θα έρθουν πιο κοντά σε εμά και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι θα επιθυμούσαμε. Ή λοιπόν θα προχωρήσουμε με τις δικές μας ε, τις δυνάμεις και τα στρατεύματά μας και αυτό ε, δεν νομίζω ότι μας αρέσει πάρα πολύ ή να βοηθήσουμε τους ίδιους Αφρικανούς να λύσουν τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ, Μιχαήλ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε και εδώ ε, και εσείς παρόντες να απαντήσετε σε ερωτήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο, πάρτε μια ανάσα πρώτα όμως, αφού μάλιστα στάσατε. ο κύριος Νάρτ. Άκουσα μια σειρά από κριτήρια ε, που αξιολογούν το λόγο για τον οποίο δεν λειτουργεί η άψα, που όντως δεν λειτουργεί. Αλλά το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τις δικές μας κυρώσεις ή με ε, τις ε, ένοπλες ομάδες. Ο κόσμος δεν σκοτώνεται και για πλάκα, ούτε για διασκέδαση, ούτε επειδή οι φυλές ε, τσακώνονται μεταξύ τους είναι πολιτιστικό. Όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, για να ζήσουν σκοτώνονται και σκοτώνουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ε, ε, τη δημοσιογράφοι και πολιτικοί και τα λοιπά, παρόλα αυτά κάνουν λόγο για ε, διαφυλετικές συγκρούσεις, αλλά κανείς δεν έχει πάει εκεί. Εγώ πήγα στον Ταρφούρ, υπήρχε πείνα. Υπήρχε έλλειψη γης. το οποίο οδήγησε στα άκρα ε, τους τοπικούς πληθυσμούς, να επιτίθεται δηλαδή σε άλλες φυλές. Δεν ήταν ε, λοιπόν ε, πόλεμος μεταξύ πολιτισμών. Πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη βοήθεια σε αυτές ε, τις δομές. Να σας μιλήσω για ένα κράτος πάρα πολύ ισχυρό και εύρωστο που είναι το Τσάντ. Είναι και υπερδιεφθαρμένη η διοίκηση εκεί, άρα είναι τεράστια η ευάλωτη κατάσταση έχω βαρεθεί να λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η Λιβύη. Το πρόβλημα είναι η μέρα που θα εκραγεί το Τσάντ και θα φτάσει σε Κονγκό, Μαυριτανία ή ε, στην ε, ε, Ερυθρά θάλασσα, όλη αυτή η θάλασσα των όπλων που υπάρχουν στην Νότια Λιβύη. Αυτή τη στιγμή μας σώζει το Τσάντ, γιατί ο στρατός τους είναι πάρα πολύ ισχυρός, αλλά βασίζεται σε μια μικρή φυλή ενός υπερδιεφθαρμένου προέδρου, ο οποίος έχει βάλει ε, να κυβερνάει φυλή του, την οποία ε, όλοι μισούν. Και σήμερα εδώ και 15 μέρες ε, γίνονται τρομερές μάχες ανάμεσα σε επίλεκτες ε, μονάδες ασφαλείας του Τσάτ που διευθύνει ο Μαχάματ Ιντρίς, που τον λένε το ψευδόνυμο του Κάκα, ε, ο γιος του Προέδρου ε, και έχει και κάτι φιλάρχους ε, που τσακώνονται με τη συγκεκριμένη αυτή δομή τη στρατιωτική. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το δει αύριο. Είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε. Γιατί νομίζουμε ότι το Τσάντ είναι μια χώρα ε, σταθερή και ο στρατός είναι παραδεκτός και μπορεί να ε, δράσει στο Μάλι και στο Νίγηρα και παντού, που δεν μπορεί να κάνει κανένας αφρικανικός στρατός και είναι ψέμα. Το πρόβλημα είναι οικονομικές και ε, κοινωνικές συνθήκες και ποιες δίκες είναι αυτές. Γιατί υπάρχει και άλλη χώρα που είναι πολύ σταθερή, πάρα πολύ σταθερή, η Μπουρκίνα Φάσο, που έχει πολύ μικρό στρατό, αλλά έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς στο Μάλι, αφού στείλαμε δεκάδες εκατομμύρια ε, ευρώ για να εκπαιδεύσουμε χωρίς όπλα τον κόσμο εκεί και δεν δίνουμε όπλα και τους ε, ε, εκπαιδεύουμε για να αμήνονται. Και αν δεν υπήρχε το Μπαρκάν και η Μινούσμα, θα ήταν στον Παμάκο οι τρομοκράτες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί δεν καταφέραμε να, κάνουμε, να φτιάξουμε ούτε ένα λόχο επιχειρησιακό. Λόχο. 120 άνδρες είναι σε πέντε χρόνια. Το πρόβλημα είναι ποιου συνομιλητές έχουμε εκεί και τι κάνουμε εκεί πέρα. Το πρόβλημα δεν είναι να στέλνουμε λεφτά, να πληρώνουμε δομές. Η οργάνωση Αφρικανικής Ενότητας ο Μούσα Φάκη είναι επικεφαλής και τον ξέρω πάνω από 35 χρόνια. Εσείς γνωρίζετε ποιος είναι ο γιος του Μούσα Φάκη. Ο γιος του είναι ένας εγκληματίας ο οποίος με πέντε συντρόφους ε, μέρες ολόκληρες βίαζαν μια ε, μικρή από το τσάτ και το βγάλαν και στο δίκτυο. Και αυτή η κοπέλα ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε πόσες μέρες ο Μούσα πήγε φυλακή, ούτε μισή μέρα. Για ποιο λόγο, γιατί είναι γιος του πατέρα του. Γενικός Γραμματέας της Αφρικανικής Ένωσης. Με αυτούς τους ανθρώπους συνεργαζόμαστε και με αυτούς τους ανθρώπους συνομιλούμε. Εγώ δεν σας μιλώ για καμιά υπερδομή, επικοδόμημα. Σας μιλώ για τους ανθρώπους και τα πεπραγμένα τους. Στο τσάτ τι γίνεται εκεί επί τόπου. Ο αδερφός του Προέδρου Λαού Σαντεμπή με ε, εταιρείε από τη Νότια Αφρική έστειλε με πυροβολισμούς ε, κάποιους ε, χρυσοθύρες στο μίσκι, αλλά στο μίσκι οι φυλές ε, εξεγείρονται και δεν τους αφήνουν να τους σκοτώνουν και καταστρέφουν το στρατό του Ντρίστιμπη. και στο, το τσάτ θα εκραγεί σε χίλια κομμάτια και τότε θα έχουμε πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα θα φτάσουν στο Κονγκό τα όπλα και στην Ερυθρά θάλασσα και στον Ατλαντικό. Και τότε τι θα κάνουμε, θα πούμε ότι χρειαζόμαστε να βρούμε μια αρχιδίκηση, στη βαρύ διοίκηση ή μια διοίκηση ε, αξιόπιστη. Γι' αυτό σας μιλάω για την Μπουρκίνα Φάσο. Τι, τι πρόβλημα έχει ο Ρόκα Μπορέ, που είναι και καλός φίλος και σοβαρός άνθρωπος, ότι στο Μάλι δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Και η Φιλίπ Πελ που ποτέ δεν έχει εξεγερθεί, έχει φτιάξει μια μονάδα που μπήκε στην Πουργίνα Φάσο. Η UPOL που δεν πληρώνεται κιόλας, οι χωροφύλακε γιατί τα λεφτά ε, ε, τα κρατάνε στον Παμάκο. Οι χωροφύλακε λοιπόν που εμείς εκπαιδεύουμε πάνε και φυλάνε γελάδια και γίδια και ε, στους, στη Φιλίπ Πέλ και τελικά όμως αυτό ε, αποσταθεροποιεί και το Μάλι και τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο. Εμένα η Αφρικανική Ενότητα με φέρνει σε ένα πραγματικά διανοητικό οργασμό. Μου φαίνεται καταπληκτικό, θαυμάσιο πλάνο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ε, ουσιαστικές συνομιλίες με γνήσιους συνομιλητές. Και το ξέρω ότι πολλές φορές πρέπει να συνεργαζόμαστε με κάποιους που δεν μας αρέσουν. Εντάξει, αλλά να είναι αυθεντικοί. Ε, το πρόβλημα δεν είναι το επικοδόμημα, είναι το οικοδόμημα, η δομή η ίδια. Συμφωνώ και εγώ είμαι απεσιόδοξος, αλλά πώς μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Γιατί όταν εξακολουθούμε να δίνουμε λεφτά σε άδειε δομές, σε διεφθαρμένες ή που τις μισεί ο ίδιος ο λαός τους, όσο και σταθερές να φαίνονται, είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο φράγμα που να συγκρατεί αυτό το τεράστιο όγκο νερού, αλλά είναι κρυστάλλινο και άμα φάει ένα πλήγμα θα σπάσει και θα μας πλημμυρίσει το νερό. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος δεν σκοτώνεται γιατί του αρέσει. Οι ε, μονάδες οι ε, τρομοκρατικές, οι τζιχαντιστικές δεν είναι ανακατέβατες. Η απόγνωση της γεννάει και θα θυμίζα σε κάποιους από τους διπλωμάτες ότι να μην πάνε μόνο στην Τζαμένα, στο Γουαγαντούγου, στην Ιαμέη και στον Παμάκο, να πάρουν τα πόδια τους και να πάνε εκεί που είναι τα προβλήματα και όχι με αυτοκίνητο με ε, σε ε, ξενοδοχείο Mercondition, σε εστιατόριο Mercondition, να δούνε τίποτα προεστούς που θα τους λένε τα ωραία πράγματα. Να πάνε να δουν πώς ζει ο κόσμος στην πραγματικότητα και τότε θα καταλάβουν ποια είναι η πραγματικότητα. Λέτε ότι έχουμε πρόβλημα επιμελητίας με τον Αφρικανικό στρατό. Δεν είναι πρόβλημα επιμελητίας, είναι ένα απόλυτο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν μονάδες στην Αφρική που δεν θέλουν να πολεμήσουν. Και αυτό είναι και φυσιολογικό, ούτε εγώ θα ήθελα. Τα λεφτά μου τα κρατάνε ε, ο λοχαγός, ο αντισυνταγματάρχης ή ο στρατηγός ή και οι τρεις μαζί και να δεν πάμε να τους δίνουμε ε, όλους τους ασυρμάτους που χρειάζονται και όλο το υλικό για να φτάσεις κάπου πρέπει να έχεις πειθαρχία και δεν υπάρχει αυτό στο στρατό και στο Κονγκό και παντού. Όσο καλοπληρωμένη και να είναι η μονάδα ε, και ε, η μηνυσκότητα των Ηνωμένων Εθνών που είναι το σκάνδαλο, τι γίνεται στην Κεντρική Αφρική επειδή δεν δίνουμε ε, χρήματα όπλα μάλλον τα δίνουν οι Ρώσοι και οι Ρώσοι με πολύ λιγότερα λεφτά παίρνουν τη μερίδα του λέοντος στην Κεντρική Αφρική και τι πταίει, ε, πταίει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δόξα τω Θεώ η Μέρκελ και ο Μακρόν κατάλαβαν ότι έχει έρθει η ώρα να βγούμε από τη μεταφυσική και τον κόσμο της και να έρθουμε στην πραγματικότητα, να προσγειωθούμε. Και σας το λέω ειλικρινά, θα πετάμε λεφτά από το παράθυρο και θα συνεχίζουμε για υπερδομές για να φτάσουμε με όλα αυτά τα λεφτά στην απόλυτη φτώχεια. Γιατί χωρίς τον Μπαρκάν που είναι οι γαλλικές μονάδες και χωρίς τη Σιέρα Λεόνε ε, που έχουμε ε, μισθοφόρους, executive outcomes, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν τίποτα, γιατί δεν έχει ούτε δυνατότητα, ε, ούτε ικανότητα, αλλά είναι μια καταπληκτική μπίζνα για τους διοικητικούς υπαλλήλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που έχουν ε, πολύ βαθιές γνώσεις για το τι ακριβώς ε, διαδραματίζεται στην Αφρικανική Ένωση και σε μεμονωμένες χώρες. Θα ήθελα τώρα πάρα πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα που τέθησαν επιτάπητος ε, και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πολύ καλά και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί αν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που θέλετε να πείτε ε, πριν δώσω το λόγο στον ε, παρακαθήμενό μου για να απαντήσει στις ερωτήσεις, μπορούμε βεβαίω αν θέλετε να συμπληρώσουμε και με άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φυσικά και σα ευχαριστούμε και για το Ελληνικό Συνέδριο. Ε, και εμείς ε, συμφωνούμε με τις ε, συστάσεις και έχουμε αρχίσει να τις υλοποιούμε. Θα ήθελα ενδεχομένω να επισημάνω ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι ως προς τα όσα έχουν ε, επιτευχθεί από την άψα και από το Ελληνικό Συνέδριο. Και η ανεξάρτητη έκθεση του 2016 από το Ινστιτούτο ε, Μελετών Ειρήνης και Ασφάλειας προέκυψε το 75% των ε, παρεμβάσεων πρόληψης ε, συγκρούσεων θεωρήθηκαν επιτυχής ή μερικώς επιτυχής. Το 2016 αυτό. 86% των παρεμβάσεων άψα θεωρήθηκαν μέσης ή ανώτερης ποιότητας από το ίδιο Ινστιτούτο. Και θα θέλαμε να επισημάνουμε και την διασύνδεση και την ανάγκη για οικονομική βιωσιμότητα της Αφρικανικής Ένωσης. Συμφωνούμε σε αυτό και μάλιστα εμείς ε, διαδραματίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη ε, των επιτροπών της Ευρωκοινικής Ένωσης για να κινηθούν προς ε, την έκθεση για το σχέδιο Καμπερούκα. Ιδίω ό,τι αφορά την ιδέα ανάπτυξης του φόρου 0,2% στις εισαγωγές. Αν δείτε το 2016, και το επιχειρησιακό κόστος. Τα κράτη της Αφρικανικής Ένωσης κάλυπταν μόλις 30% του, των λειτουργικών δαπανών. Αν δείτε πώς έχουν τα πράγματα το 2018, πλέον αυτό έχει ανέβει στο 75%. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη έχει μειωθεί το δικό μας μερίδιο στην κάλυψη αυτών των δαπανών. Οπότε, ήδη μειώνεται αυτή η συνεισφορά, όπως έχει συστήσει το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα, κατά πόσο πρέπει να στεκόμαστε και να βασιζόμαστε στα αποτελέσματα, συμφωνούμε πλήρω με αυτή την προσέγγιση και σύσταση. Πρέπει να βελτιωθούμε. Στην επόμενη φάση υποστήριξης ε, του άψα μαζί με την Αφρικανική Ένωση. Το επισημαίνουμε αυτό και οι δύο θα πρέπει να επικεντρωθούν σε, σε έναν αριθμό μειωμένων προτεραιοτήτων και να θέσουν πολύ συγκεκριμένου στόχου και δείκτε που θα μας επιτρέψουν να μετρήσουμε τα αποτελέσματα και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Όλα αυτά έχουν ήδη ενταχθεί στις συζητήσεις μας για την προετοιμασία του προγράμματος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς ε, να πω ότι πράγματι ε, υπάρχει ανάγκη η μείωση των καθυστερήσεων και της αναδρομικής ισχύω. Ίσως ε, να υπάρχει βέβαια ένα δύσκολο πλαίσιο στο οποίο ε, ενεργεί αυτή τη στιγμή το ΑΠΣΑ εξαιτία και των ε, θεσμικών αδυναμιών των ομολόγων μας. Όμως έχουμε αναλάβει δράση, ιδίω σε σχέση με πριν από δύο χρόνια και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για να ε, ενισχύσουμε και την οικονομική στήριξη της Αφρικανικής Ένωσης για να λειτουργούν και αυτοί καλύτερα σε ό,τι αφορά και την ποιότητα των εκθέσεων, γιατί η κακή ποιότητα αυτών των εγγράφων είναι η απαρχή και η αιτία των καθυστερήσεων που έχουμε στη συνέχεια στις συμβάσεις. Και γι' αυτό το λόγο και από πλευράς μας έχουμε αυξήσει τις ικανότητές μας για την ε, ε, επίλυση αυτών των ζητημάτων. Θα μείνω εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περέιρα. Λοιπόν, ε, ακούσατε πολλά σχόλια και παρατηρήσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους συναδέλφους μου που επεσήμεναν τις δυσκολίες που υπάρχουν και ο Χαβιέ και ο Μίκαλ ανέφεραν ε, συγκεκριμένα ζητήματα. Ακούμε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους ε, που πήραν το λόγο προηγουμένω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βεβαίω. Δεν θέλω βέβαια να ξεφύγω από ε, το αντικείμενο της έκθεσης. Να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα τον κύριο Νάρτ, γιατί αυτό που αναφέρατε πρέπει κάπως να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της στρατηγικής. για να ζητήσουμε την ανάληψη ευθυνών από τους δωρητές. Αυτό που κάνουμε και κατά την κατάρτιση της ε, έκθεσης. Να δούμε λοιπόν τι είναι εφικτό στην πράξη και τι όχι. Βασική μας σύσταση γι' αυτό ήταν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την αφρικανική πλευρά να αναλάμουν τις βασικές οικονομικές τους ε, ευθύνες και υποχρεώσεις, γιατί έτσι δείχνουν και τη βούλησή τους, ε, την οποία έχουν διακηρύξει πριν από 15 χρόνια. Ότι για, την, για τα αφρικανικά προβλήματα πρέπει να υπάρχουν αφρικανικές λύσεις και ούτω καθεξής. Διαφορετικά μπορεί να έχουμε ε, πολύ καλούς οδικούς χάρτες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Και χαίρομαι που υπήρχε καλός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο μέλλον θα φανεί ότι η επανεστίαση στη πραγματική οικοδόμηση ικανοτήτων για την αφρικανική ασφάλεια είτε σε παναφρικανικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, όχι απλά η κάλυψη των δαπανών και του κόστου. Τι μορφή θα λάβει η στρατηγική θα φανεί στο μέλλον, αλλά χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπα και προηγουμένως, ήδη έχουν περάσει στη φάση της υλοποίηση. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική τη ε, μορφή στη συνέχεια. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Αλλά και αυτό που είπε ο κύριος Γκάλερ είναι σαφές, ότι υπάρχει μια τέτοια στρατηγική σύγχυση. Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να επενδύσουμε ε, σε αυτή την οικοδόμηση ικανοτήτων, σε αφρικανικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί και οι περιφέρειες διαφέρουν, ε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα όμως γιατί τότε μπορούμε να δούμε πραγματικά την απόδοση και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε βιώσιμα αποτελέσματα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάρτς. Ακούσαμε την απάντηση και βέβαια και τα σχόλια του κυρίου Περέιρα. Έχετε άλλα σχόλια, παρατηρήσεις, συνάδελφοι, επιθυμεί κανείς να πάρει το λόγο. Ο Μιχαήλ Γκάλε. Σε ε, επίπεδο αφρικανικών κρατών, ε, διοικητικών και κοινοβουλευτικών μπορείτε να στείλετε σε όσους περισσότερους μπορείτε αυτή την έκθεσή σας να ε, διαδοθεί όσο γίνεται περισσότερο στην Αφρική για να πυροδοτήσει και κάποιες επικοδομητικές συζητήσεις. Ε, μια σύντομη απάντηση ο κύριος Πάρτς. Ε, ε κοιτάξτε, ε, ο τύπος και τα μέσα ενημέρωσης κάλυψαν ευρέως το γεγονός στην Αφρική και εφημερίδες και τηλεόραση και τα επιγραμμικά μέσα κτλ. Οπότε, αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, ευχαριστώ τους συναδέλφους για την παρουσία τους και τον κύριο Περέρα και τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήρθαν στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τον κύριο Πάρς του Ελεκτικού Συνεδρίου που ήρθε ε, εδώ για να μας παρουσιάσει την ειδική τους έκθεση. Το εκτιμούμε τα μάλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τούτων των όλων λεχθέντων ολοκληρώσαμε τις ε, σημερινές μας εργασίες και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9. Και έχετε και τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ.